Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε γιατί βλέπω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι που ασχολούνται με το πρώτο θέμα, τον τελωνιακό κώδικα, είναι εδώ, είναι εδώ και η συγγήτρια. Να σας κάνω κάποιες ε, αρχικές ανακοινώσεις. Καταρχάς, να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Ωραία, εγκρίνεται, σας ευχαριστώ. Βλέπετε ότι έχουμε μια ωραία αίθουσα, μπαίνει και ο ήλιο. Επομένω, μπορούμε να βγάλουμε και καλύτερε φωτογραφίε στο διαδίκτυο, γιατί η συνεδρία μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Θα ψηφίσουμε και την έκθεση για τι δημόσιε συμβάσει. Προτείναμε μια αναβολή κατά ένα μήνα, τρει εβδομάδε είναι στην πραγματικότητα, διότι οι συγητές και οι σκιώδει συγητές έχουν ακόμα πολλή δουλειά. Είναι πολύ περίπλοκο το κείμενο και έχει και ε, πάρα πολλές ε, τροπολογίες και ε, συμφωνήσαμε ότι καλύτερα ήταν να ολοκληρώσει αυτή τη δουλειά για να έχουμε και μια κάποια ποιότητα και να έχουμε στη συνέχεια μια ισχυρή ψηφοφορία που θα βρει και σύμφωνα τα περισσότερα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Επιτροπής μας συγγνώμη, για να έχουμε μια κοινή θέση. Θα καθυστερήσουμε λοιπόν το χρονοδιάγραμμα για να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία. Στις 18 Δεκεμβρίου λοιπόν θα έχουμε τις ε, δημόσιες συμβάσεις και το χρόνο το οποίο θα αφήσουμε ε, θα τον αξιοποιήσουμε κάνοντας μια συνεδρία και κλεισμένων των θυρών για να συζητήσουμε κάποιες λεπτομέρειες από του θέατος. Να σας πω επίσης ότι έχει εκδοθεί η νέα εκδοχή του newsletter μας. Ε, οι συνάδελφοι θα πρέπει να έχουν λάβει και αντίγραφο στα γραφεία τους. Όποιος ε, δεν έχει ε, ζητήσει ήδη να λαμβάνει το newsletter μπορείτε να το ζητήσετε και να το παίρνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο κάθε μήνα. Όπως σας είπα και προηγουμένως μεταδίδεται και μέσω, του, μέσω web streaming και συνεδρίαση. Επίσης να σας πω ότι η Επιτροπή έχει πλέον λογαριασμό στο Twitter. Το ήξερα ότι θα σας χαροποιήσει αυτή η είδηση. Έχουμε λοιπόν δίαιση ε, EP κάτω παύλα single market όλα σε μία λέξη. Θα σας το στείλουμε βέβαια κιόλα το hashtag. Και εκεί λοιπόν θα ε, βλέπετε σημειώσεις για τα, τη συνεδρίαση, ε, των συνεδριάσεών μας, ε, θέματα για την ημερήσια διάταξη και επίσης τις διαδικασίες. Μπορείτε να βλέπετε λοιπόν και για τις διαδικασίες ζωντανά στο Twitter και τα μέλη τα οποία είναι δραστήρια στο Twitter μπορούν να προσθέσουν ένα σύνδεσμο στον, στην ε, επιτροπή μας, η EP Single Market, ε, στον λογαριασμό τους στο Twitter. Κυρία Κέλλερ, ήθελα να διευκρινίσω κάτι για το χρονοδιάγραμμα της ψηφοφορίας για τις δημόσιες συμβάσεις και να σας πω να ψηφίσουμε το πρωί στις 18 και όχι το απόγευμα, Θα το εξετάσουμε, λέει ο Πρόεδρος. Ε, έχουμε πάρα πολλές ψηφοφορίες και επίσης τον Ιανουάριο ε, θα έχουν πολλή δουλειά και για τα Χριστούγεννα γιατί θα ε, ψηφίσουμε και τις δημοσίες συμβάσεις και την αναγνώρι... αμοιβαία αναγνώριση ε, επαγγελματικών προσόντων ε, και τις κοινοφελείς υπηρεσίε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα είναι μαραθώνια η ψηφοφορία και μπορείτε να τα γράφετε και στο Twitter όσο θα ψηφίζουμε. Έχετε επίση τα πρακτικά τη συνεδρίαση τη 5η και 6η Νοεμβρίου. Εάν δεν υπάρξουν ενστάσει μέχρι το πέρα τη συνεδρίαση, θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Και τώρα να περάσουμε στο πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη για τον εξυγχρονισμό του τελωνιακού κώδικα της Ένωσης, την αναδιατύπωση του συγκεκριμένου κανονισμού. Πρόκειται για μια περίπλοκη και δύσκολη ε, πρόταση. Η κυρία Λεγκρίπ ε, είναι πολύ δραστηρία, το ίδιο και σκιώδης συγητές. Ε, θα μας πει λοιπόν πού ακριβώς βρισκόμαστε. Έχουμε περίπου 250 τροπολογίες. Είναι και η κυρία Ράπτη εκ μέρους των σοσιαλιστών, σκιώδης συγητρία. Ο, ο κύριος Βάντερκαμπ, ο κύριος Σμιτ είναι εδώ, εκ μέρους των φιλελευθέρων. Συγγνώμη, ο κύριος Βαντερκάμπ είναι από την εβδομάδα, ο κύριος Χατζημαρκάκης μόλις ήρθε, η κυρία Μακλάρκινγκ μιλάει εξ μέρους του κύριου Μπίλεν και η κυρία Σαλβίνη δεν είναι εδώ ακόμα. Να προχωρήσουμε λοιπόν. Να καλωσορίσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Ζαμισελ Γκράφ, ο οποίος είναι επικεφαλής ε, του τμήματος για τον ε, τελωνιακό κώδικα. Θα μιλήσει λοιπόν με τους εισηγητές και οποιονδήποτε βέβαια θέλει να συμμετάχει στη ε, συζήτηση. Κύριε Λεγκρίπ, να σας δώσω το λόγο για να μας παρουσιάσετε τα της πρότασης. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και ευχαριστώ που θα συζητήσουμε πάλι την τροπολογία με, όσον αφορά την ανασύσταση του ελληνικού κώδικα. Ε, της Ένωσης. Οι τρεις στόχοι αυτή της αναμόρφωσης, όπως παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή μας στις 26 Απριλίου, είναι πρώτον να αναβληθεί η ημερομηνία εφαρμογή που προβλεπόταν ε, στις 24 Ιανουαρίου 2013, ε, διότι ο κανονισμός του 2008 δεν θα μπορεί να τηρηθεί λόγω σημαντικών αλλαγών στο πληροφοριακό σύστημα και στην καθυστέρηση ορισμένων κρατών μελών όσον αφορά τη μετατροπή του συστήματος. Δεύτερος λόγος για αυτή την αναδιατύπωση πρέπει να προσαρμοστεί ο κώδικας με την έναξη ισχύω της συνθήκης αβώνα, ε, ποιε είναι οι πράξει ε, εφαρμογή κτλ. Ε, 92. Τρίτος στόχος, να ληφθούν υπόψη οι κανονισμοί στις, ε, του τομελεγών κανονισμών όσον αφορά τις διαδικασίες πληροφορικής. Το σχέδιο έκθεσης, το οποίο είχα την τιμή να σας παρουσιάσω στις 17 Σεπτεμβρίου, ε, θέλησα να υπάρξουν ορισμένες διατάξεις, ώστε να υπάρξει στο μέτρο του δυνατού συνένεση μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων, εμπλεκομένων του τελεινιακού κόσμου. Πρώτο θέμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή τη διαδικασία αναδιατύπωσης. Συνεπώς, η διαδικασία κατάθεσης των τροπολογιών χαρακτηρίστηκε από τους κανόνες που ισχύουν στην αναδιατύπωση μέσα στα νομοθετικά μας κείμενα. Γι' αυτό υπήρξε μια κοινή βούληση μεταξύ των σχεδόν εισηγητών και μου σε μια προσπάθεια να αλλάξουμε διατάξεις της αρχικής πρότασης Επιτροπής ακόμα και σε ορισμένα τμήματα που ονομάζονται λευκά. Θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω σε αυτή την ιδιότυπη διαδικασία διατύπωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να προβεί σε τροπολογίες ε, στις, στα γκρίζα μέρη, στα γκρίζα τμήματα, αλλά για να μπορέσει το Κοινοβούλιο να επιφέρει τροπολογίες στα λευκά τμήματα και αυτή είναι μια αρχή που πηγάζει από την Διεθνική Συμφωνία και έχει σχέση με την τεχνική αναδιατύπωση των νομικών πράξεων, τότε θα πρέπει να υπάρξει πολιτική συμφωνία, όσο το δυνατόν ευρύτερη, μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δουλέψουμε πάνω σε ορισμένα θέματα και ε, να επιτύχουμε αυτή την πολιτική συμφωνία. Ήδη άλλωστε στην πρώτη μου παρουσίαση είχα εκφράσει την επιθυμία να αλλάξουν τις μέρες διατάξεις αυτού του περίφημου λεγόμενου λευκού τμήματος. Και είχαμε την ε, συμφωνία των περισσότερων ε, σχεδόν συγητών με σκοπό να στείλουμε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα από το κοινοβούλιο μας όσον αφορά την εμβάθυνση της Τελωνιακής Ένωσης, όσον αφορά την βελτίωση, την αναβάθμιση ε, των οικονομικών, ε, του καθεστώτος των οικονομικών φορέων, αλλά και για μεγαλύτερη απλούστευση και για ασφάλεια, μεγαλύτερη ασφάλεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους χιώδεις που με βοήθησαν και που θέλησαν να συνυπογράψουν κοινέ τροπολογίες ή που τις ενέκριναν. Προχωρήσαμε λοιπόν με τους χιώδεις πάνω σε δύο μείζωνα θέματα την προσωρινή κατάθεση. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα λεγόμενο λευκό τμήμα της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. Θελήσαμε να καταθέσουμε τροπολογίες που θα επιτρέπουν να επανέλθουμε στο πνεύμα του εξυγχρονισμένου Ελληνικού κώδικα και λαμβάνοντας υπόψη αυτό το ε, προσωρινό καθεστώς σύμφωνα με τα όσα μας είχε πει η Κομισιόν στο κείμενό της. Επισημοποιήσαμε τις προτάσεις μας όσον αφορά τις προσωρινές καταθέσεις και εδώ έχουμε ορισμένε τροπολογίε και ελπίζουμε ότι οι θέσει μα θα γίνουν δεκτές από τα άλλα θεσμικά όργανα. Αλλά οπωσδήποτε ε, θέλουμε να ακούσουμε πάνω σε αυτό το θέμα της προσωρινής κατάθεσης ε, της ε, επιτροπή της Επιτροπής και του Συμβουλίου, αν το επιθυμεί, ώστε να γνωρίζουμε ποια είναι η απόψή τους. Ένα δεύτερο μείζον θέμα μετά από την προσωρινή κατάθεση, η αναβάθμιση ε, της ιδιότητας ε, των αναγνωρισμένων ε, φορέων. Δηλαδή αυτό που θέλουμε είναι το καθεστώς αυτών των αναγνωρισμένων φορέων να γίνει το μέσο για την απλούστευση για τους οικονομικούς μας φορείς. Είναι πρωταρχική σημασία οι φορείς οι οποίοι προβαίνουν στις αναδιατυπώσεις και τα τις απαραίτητες διατυπώσεις ε, που είναι μακροχρόνιες και κοστίζουν πολύ, είναι σημαντικό, επαναλαμβάνω, αυτά τα άτομα να μπορούν να έχουν αυτό το καθεστώς, την ιδιότητα και να απολαμβάνουν πραγματικών και συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων. Η αναβάθμιση αυτής της του, τους, θέσεώ τους, θα πρέπει να τους επιτρέψει να πείσουν για ε, το ενδιαφέρον που παρουσιάζει αυτό το νέο καθεστώς. Και μαζί καταθέσαμε τουλάχιστον σε ένα πνεύμα κοινό περίπου πέντε τροπολογίες για να αναβαθμίσουμε την θέση αυτών των φορέων. Όσον αφορά λοιπόν πάντοτε τα λεγόμενα λευκά τμήματα του αρχικού κειμένου, όπου μόνον εμείς οι σκιώδει συγητέ, οι και, και άλλα μέλη τη Επιτροπής μας θελήσαν να καταθέσουν τροπολογίες, υπάρχουν αρκετοί, θα έλεγα, Υπάρχουν αρκετές τροπολογίες, τις οποίες εξετάσαμε εντάχει στη συνεδρίαση των σχεδόν εισηγητών και μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν μεγάλες αντιρρήσεις από πλευράς ε, εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες θα υποστηριχθούν, αλλά στο παρόν στάδιο δεν θελήσαμε να τις σταματήσουμε, να τις μπλοκάρουμε και δεν θα έχουμε αντίθεση αν χρειαστεί να συζητηθούν. Γι' αυτό το λόγο, κύριε Πρόεδρε, ως εισηγήτρια πάντοτε στα, για τα λεγόμενα λευκά τμήματα, σας κυκλοφορήσαμε ένα κατάλογο τροπολογιών που καταθέσαμε εμείς και οι στιώδεις ηγητές και τα άλλα μέλη της Επιτροπής μας, που ίσως σας φανούν πολλά, γιατί τελικά οι τροπολογίες είναι 71 τροπολογίες, όσον αφορά δηλαδή την προσωρινή κατάθεση, αλλά και βελτίωση του καθεστώτος των αναγνωρισμένων φορέων, αλλά και για άλλα θέματα που θέλησαν να συζητήσουν οι συναδελφοί μας. Και θα δούμε πώς μπορούν να διατηρηθούν, να παραμείνουν αυτές οι τροπολογίες στη συζήτηση. Γενικότερα τώρα, ως προς τα διάφορα θέματα που εφήγησαν στις διάφορες τροπολογίες που κατατέθηκαν, είτε πρόκειται για τροπολογίες που κατέθεσαν σκιώδεις συγητές, είτε από άλλα μέλη της Επιτροπής μας. Και εδώ, αν θέλετε, συσσωρεύω τις τροπολογίες για τα λευκά τμήματα και τις πολλές τροπολογίες για τα γκρίζα τμήματα του κειμένου, επειδή τα δεύτερα θα μπορούσαν να τροποποιηθούν, τα θέματα είναι τα εξής όπως είπα, αναβάθμιση της θέσεως, της ιδιότητας των αναγνωρισμένων φορέα, ε, πέραν από τις διάφορες τροπολογίες που ανέφερα, που κατατέθηκαν από πολλά μέλη, αλλά που γενικά η πλειοψηφία εξ αυτών τουλάχιστον ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή ε, οι κοινέ μα τροπολογίε των εισηγητών και σχεδόν εισηγητών, όπω είπα στην έκθεσή μου. Όλε οι τροπολογίε λοιπόν έχουν ω αντικείμενο να καταστεί αυτό το καθεστώ πιο ελκυστικό πιο λειτουργικό προκειμένου να υπάρχουν σημαντικά συγκεκριμένα πλεονεκτήματα. Υπάρχουν 12 περίπου τροπολογίε που κατατέθησαν από του μεν και από του δε, που ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση και έχουν την ίδια φιλοσοφία. Επίσης, ορισμένοι συναδελφοί μα θέλησαν, όπως έκανα και εγώ στο σχέδιο έκθεσή μου, να περιλάβουν στο βασικό κείμενο τις διατάξεις που θεωρούν ουσιαστικές. Το είχα αναφέρει πρωτήτερα και μάλιστα στο σχέδιο εκθεσή μου, αν θέλετε, περιέλαβα και πάλι διατάξεις που θεωρώ ουσιαστικές ε, από το βασικό κείμενο και ορισμένοι από τους συναδέλφους μας πάλι ε, συμφωνούν και για αυτό το λόγο ανέλαβαν σχετικές πρωτοβουλίες. Γνωρίζω βεβαίως ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί προκειμένου το τελικό κείμενο να μην είναι πολύ βαρύ ούτε πολύ μακρύ και γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε, να εξασφαλίζουμε συνοχή, να είναι βανάγνωστο το κείμενο, να είναι απλό και γι' αυτό θα προσπαθήσω να λάβω υπόψη τις τροπολογίες που έχουν ως αντικείμενο ε, να ε, γίνει το κείμενο πιο σαφές, πιο απλό και πιο βανάγνωστο. Άλλο, άλλο θέμα, ορισμένοι συνάδελφοι θέλουν απλούστευση ορισμένων διαδικασιών ε, σύμφωνα με την αρχική συνοπτική δήλωση και μια τελική δήλωση. Οι περισσότερες ε, τροπολογίες που κατατέθηκαν έχουν σαν αντικείμενο επιτρέψουν στους οικονομικούς φορείς ή στους ε, αναγνωρισμένους φορείς να εξαιρεθούν από ορισμένε και υποχρεώσεις. Δεν έχω καταρχήν αντίρρηση ως προς αυτό το σκοπό, τον οποίο συμμερίζομαι στις γενικές του γραμμές. Απλά πρέπει να δούμε με μεγάλη προσοχή αυτή την επιθυμία, δηλαδή η... να αρθούν ορισμένες υποχρεώσεις ή να περιοριστούν. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αποκλειστούν όλα. Θα πρέπει να βρούμε μία ισορροπία ε, στην Τελωνιακή Ένωση διότι ρόλος μας είναι η προστασία, η εγγύηση της ασφάλειας και συνεπώς οι διάφοροι έλεγχοι, οι διάφορες ε, διατυπώσεις πρέπει να διατηρηθούν. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία όταν μιλάμε για απλούστευση. Ναι, απλούστευση, αλλά εγγύηση ασφάλειας, τήρησης κανόνων όσον αφορά πάντοτε την ασφάλεια. Και άλλα θέματα θίγονται στις τροπολογίες που κατατέθηκαν από διάφορες ομάδες που θα πρέπει πάλι να συζητήσουμε εις βάθος, κυρίως μεταξύ εισηγητών και σχεδόν εισηγητών, αναφέρουμε κυρίως τη δυνατότητα να έρθει υποχρέωση ε, για έναν φορέα αναγνωρισμένο να παρουσιάζει διατυπώ όταν είναι εγκατεστημένο σε ένα κράτο μέλο τη Ένωση. Εδώ πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στι θέσει ε, των μελών που θέλουν την απαγόρευση, δηλαδή την άρση υποχρέωση, και εκείνων που επιθυμούν να ενσωματωθούν με συγκεκριμένο τρόπο και αυστηρό. Επόμενο θέμα. Οι κανόνε προέλευση. Ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ορισμένε τροπολογίε, σημαντικέ, ενδιαφέρουσε κατατέθηκαν πάνω σε αυτό το θέμα των κανόνων προέλευσης, θα προσπαθήσω να προτείνω μια συμβιβαστική τροπολογία σύμφωνα με τη γενική φιλοσοφία των διαφόρων τροπολογιών που θα επιτρέπει, ελπίζω, εάν υιοθετηθεί και στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο, να έχουν μια ισχυρή θέση και ενιαία. Μιλάμε εδώ για τους κανόνες απόκτησης καταγωγής ε, τώρα, ποια είναι η τελωνιακή αξία και ο προσδιορισμός. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν άφησε διάφορους του συναδέλφους επ' αυτού του θέματος, όπως και για τους κανόνες από τις καταγωγής, δηλαδή ο προσδιορισμός της τελωνιακής αξίας, ε, χρειάζεται ακόμη να γίνει δουλειά για να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια συμβαστική τροπολογία που ε, θα συγκεντρώνει την πλειοψηφία μας. Τώρα, η, όσον αφορά τις παρεκκλήσεις του άρθρου 6, είναι το άρθρο το, σύμφωνα με το οποίο η ηλεκτρονική βοήθεια θα πρέπει να είναι, τα ηλεκτρονικά μέσα θα πρέπει να είναι η διαδικασία για κάθε ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ε, τελωνιακών αρχών, οικονομικών φορέων και τελωνιακών αρχών. Αυτή η αρχή έχει σαν αντικείμενο διευκολύνει την ε, αλληλενέργεια, την ε, συνεργασία μεταξύ των αλλά και ασφαλίζει την ασφάλεια της ανταλλαγής εμπορευμάτων στην επικράτειά μας. Συνεπώς και εδώ νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να βρεθεί ένας συμβιβασμό που θα επιτρέπει να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη φόρμουλα. Έρχομαι τώρα στο ευαίσθητο θέμα της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ ε, πράξεων εκχωρήσεων και πράξεων εκτέλεσης. Είναι κάτι το οποίο πρόσφατα συζητήσαμε στο Κοινοβούλιο και εδώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε συνοπτική, ε, συνεκτική και σφαιρική αντιμετώπιση, ώστε οι προνομίες και οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου μας να γίνουν σεβαστές. Φυσικά αυτό το θέμα της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ ε, πράξεων ε, κατεξιοδότηση εκτελεστικών πράξεων δεν πρέπει να μας δημιουργήσουν προβλήματα. Αλλά πιστεύω ότι κάθε θεσμικό όργανο πρέπει να καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να βρεθεί ε, ένας χώρος όπου θα συμφωνούμε με βάση ε, τη λογική ε, εφόσον η Τελωνιακή Ένωση πρέπει να είναι ο πραγματικός πυλώνας ε, της εσωτερικής αγοράς. Στο παρόν στάδιο θέλω να σας πω ότι ορισμένε τροπολογίες, κοινοβουλευτικές τροπολογίες που κατατέθηκαν είναι αντίθετες προς τη θέση η οποία θα πρέπει να είναι εκείνη του Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα της κατανομής των αρμοδιοτήτων. Δεν θέλω να τις αναφέρω στις τροπολογίες, αλλά θα έλθω σε επαφή με τους συναδέλφους που τις κατέθεσαν και να δούμε κατά πόσον είναι σκόπιμες πάντοτε προς το συμφέρον ε, και για την προστασία των προνομίων ε, του Κοινοβουλίου σα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ερχόμαστε τώρα στην τελική ευθεία των εργασιών μα στα πλαίσια τη Επιτροπής ΙΜΚΟ. Θα ήθελα με όλου του σκιώδη ηγητέ και τα άλλα μέλη τη Επιτροπή που το επιθυμούν να συνεχίσω αυτή τη, αυτό το έργο συνεργασία, ε, με ένταση, περίπλοκο έργο, αλλά πολύ ενδιαφέρον. Και σε αυτά τα πλαίσια προτείνω μια νέα συνεδρίαση των σχεδόν συγκητών να λάβει χώρα στην επόμενη ολομέλειά μας στο Στρασβούργο και θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια ημερομηνία που θα μας βρίσκει όλους σύμφωνους. Στο παρόν στάδιο θα ήθελα να σας πω ότι θα ήθελα να ακούσω τα σχόλια της Επιτροπής και του Συμβουλίου, αν έχουν βεβαίω για την πρόοδο των εργασιών μας. Καταλήγοντας, θα ήθελα να σας πω, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι αντικείμενό μας είναι να έχουμε μια πιο, ε, μια τελωνιακή ένωση που θα έχει μεγαλύτερο βάθο και θα λειτουργεί καλύτερα υπέρ τη ανταγωνιστικότητα, τη ανάπτυξη και τη απασχόληση στην Ευρώπη. Μια τελωνιακή ένωση που θα πρέπει στο μέτρο του δυνατού να περιορίσει τι διοικητικέ δυσκολίε, τη γραφειοκρατία που βαρύνουν του οικονομικού μα φορεί, διατηρώντα όμω τι εγγύσει ασφάλεια που είναι τόσο σημαντικέ για τις ανταλλαγέ στα πλαίσια της Ένωσής μας, τόσο σημαντικές επίσης για την κοινωνία μας και για την διατήρηση και την τήρηση των κανόνων της κοινωνίας μας. Η συνεργασία που επιθυμώ να συνεχίσουμε θα πρέπει να μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε μια ισχυρή θέση του Κοινοβουλίου μας. Έχουμε όλοι τον ίδιο στόχο να εμβαθύνουμε την Τελωνιακή Ένωση, διότι μια πιο αποτελεσματική Τελωνιακή Ένωση, η οποία θα λειτουργεί με αρχές πιο σύγχρονες και πιο ρεαλιστικές είναι ένα σημαντικό κρίκο για την εμβάθυνση τη εσωτερική αγορά, την οποία είμαστε όλοι τόσο προσιλωμένοι στα πλαίσια αυτή τη Επιτροπή. Well, thank you very much, Mrs. Legrip, for your... Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λεγκρίπ, διότι έχετε διαδραματίζεται καθοριστικό ρόλο σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα και καθορίζεται και σαφώ ε, κάποια θέματα τα οποία είναι ευθύνη μα λόγω τη αναδιατύπωσης του συγκεκριμένου κανονισμού. Και όπω είπατε υπάρχουν και κάποια επιπλέον τμήματα ε, τα οποία χρησιμοποιείτε προκειμένου να τροποποιήσετε κάποιε αρχέ που βρίσκονται εκτό των βασικών αλλαγών του κώδικα. Θίξατε κάποια θέματα τα οποία αποτελούν και αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να κάνουν και αυτοί αλλαγέ στο βασικό κείμενο. Αυτό είναι θέμα της οργανικής συμφωνίας μεταξύ μας. Αλλά συμφωνώ λοιπόν ότι εάν καταφέρουμε να επιφέρουμε αυτές τις αλλαγές στο βασικό κείμενο θα είναι μια ισχυρή φωνή από πλευράς μας. Να ακούσουμε λοιπόν τους κοιόδης εισηγητές. Θα ξεκινήσω με την κυρία Ράπτη. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια, την κυρία Λεγκρίπ, για την πολύ καλή δουλειά που κάνει, την πολύ δύσκολη και ευαίσθητη δουλειά που κάνει. Αισθάνομαι την ανάγκη να το υπογραμμίσω αυτό. Ε, περιέγραψε τα ζητήματα με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια και πάρα πολύ μεγάλη καθαρότητα. Αυτό με διευκολύνει γιατί θα είμαι εγώ πολύ σύντομη, κύριε Πρόεδρε. Ε, λοιπόν, στο ζήτημα της προσωρινής εναπόθεσης. Δεν θα αναφερθώ διεξοδικά, διότι η το ανέλησε επαρκώς, θα έλεγα κάτι παραπάνω από επαρκώς. Ε, καταθέσαμε και μαζί της ε, τροπολογίες και μαζί με άλλους συναδέλφους των άλλων ομάδων και πραγματικά πιστεύουμε πως οι, οι, οι, οι τροπολογίες αυτές θα βοηθήσουν στο να απλοποιήσουμε και να διευκολύνουμε τις διαδικασίες με τρόπο που να είναι και αποτελεσματικός αλλά και ασφαλής έχουν σημασία πολύ μεγάλη και τα δύο αυτά ζητήματα. Το άλλο ζήτημα είναι ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας. Εδώ τίθεται ένα ζήτημα με τις πράξεις εξουσιοδότηση. Εφόσον η συγγήτρια ζητά με τροπολογίες της τα βασικά θέματα που αφορούν το καθεστώς του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα να ρυθμίζονται στο βασικό σώμα του κώδικα, όπως ισχύει και με τον κώδικα που βρίσκεται εν ισχύ, νομίζω πως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι ακριβώς θα αναθέσουμε στην Επιτροπή να προσδιορίζει. Είναι ένα θέμα αυτό του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα οικονομική περίοδο. Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες, όχι για λόγο ε, για λόγους προστατευτισμού, αλλά κυρίως για να προστατεύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το διευκρινίζω αυτό για να μην δημιουργηθεί κάποια παρεξήγηση. Δεν έχω στο μυαλό μου τον, ε, τον προστατευτισμό, επαναλαμβάνω, έχω στο μυαλό μου τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, πηγαίνουμε στο θέμα της α, ηλεκτρονικής εποχής για τα τελωνία. Ε, είναι κάτι που νομίζω ότι το θέλουμε, νομίζω ότι το χρειαζόμαστε και θα είναι για καλό όλων. Ωστόσο, ε, εκτιμώ ότι θα πρέπει να είναι δυνατόν οι διασαφήσεις να κατατίθενται, αλλά ταυτοχρόνως να μπορούν και να διατίθενται ηλεκτρονικά. Να μην μείνουμε δηλαδή μόνο στο ότι καταθέτω τη διασάφηση, τελεία, μένω εκεί. Καταθέτουμε τις διασαφίσεις αλλά μπορούμε ταυτοχρόνως να τις διαθέτουμε και ηλεκτρονικά. Ε, ζητάμε επίσης να εξειδικευτούν οι περιπτώσεις στις οποίες έρεται η υποχρέωση να υποβάλουν συμπληρωματική διασάφιση. Ε, τέλος, ζητάμε να διευκρινιστεί στο σώμα του κώδικα ε, άλλη μια περίπτωση για την οποία οι διασαφιστές δεν είναι υποχρεωμένοι να είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για τις χώρες οι οποίες συνορεύουν με, τον, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτοχρόνως χρησιμοποιούν το ίδιο σύστημα στα τελωνία. Εδώ βάζω μια τελεία. Ε, έχουμε ακόμη δουλειά μπροστά μας, πολλή δουλειά. Ε, όπως και η συγγήτρια είπε, υπάρχουν οι συμφωνίες σε γενικό πλαίσιο, αλλά υπάρχουν εκείνες οι μικρές λεπτομέρειες, ε, εκείνα τα μικρά σημεία, αλλά πολύ σημαντικά, στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, αλλά νομίζω ότι στο τέλος θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία και ε, νομίζω ότι θα προχωρήσουμε με τον, πλέον, με τον πλέον αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά την κυρία Λεγκρίπ και τους υπόλοιπου σκιώδη με τους οποίους συνεργαζόμαστε και ευχαριστώ και τον Πρόεδρο που ε, μας βοηθά σε αυτό το πολύ πολύ δύσκολο θέμα. Uh, ευχαριστώ κύριε Χατζη Ε, θα ήθελα απλώς να ζητήσω συγγνώμη, διότι θα φύγω αυτή τη στιγμή επειδή έχω μία άλλη έκθεση που υποστηρίζω σε διπλανή αίθουσα και θα επανέλθω. Το, το λέω αυτό μη θεωρηθεί ότι ε, δεν με ενδιαφέρει από εδώ και πέρα η διαδικασία. Με ενδιαφέρει, αλλά όπως ξέρετε πρέπει να κάνω παράλληλα και μια άλλη δουλειά. Uh, Βεβαίως. Θα σας ξανακαλωσορίσουμε. Κύριε Μαρκάκη για τον κύριο Σμίτ. Ναι, για τον Όλε Σμιτ που θέλει να ευχαριστήσει την εισηγήτρια και τους σκιώδης για την καλή προετοιμασία και τις προτάσεις για να τροποποιήσουν το λευκό τμήμα που αναφέρθηκε. Το Κοινοβούλιο σε αυτό το λευκό κομμάτι μπορεί να ε, βαδίσει στα σίγουρα και να ωφελήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλε Σμιτ όμως δεν γνωρίζει σε σχέση με την κατάργηση της ε, προσωρινής αναπόθεση στο άρθρο 134. Η εναρμόνιση χρειάζεται για να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη-μέλη θα φτάσουν σε ικανοποιητικό επίπεδο τελωνιακής εποπτείας, αλλά ο συνάδελφος Όλεο Σμιτ θέλει να τονίσει ότι η Κομισιόν θα πρέπει να μπορεί να χορηγεί εξαιρέσεις ε, στα κράτη-μέλη για να ελέγχει τροποποιήσεις και απλοποιήσεις στην εφαρμογή της τελωνιακής νομοθεσίας. Τέλος, νέες τεχνικές και τεχνολογίες θα ωφελήσουν όλα τα κράτη-μέλη. Η τελωνιακή αξία είναι πολύ σημαντική για να καθοριστεί το τελωνιακό χρέος και έχει άμεση επίπτωση στους δασμούς που εισπράττονται και στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ε, θα πρέπει να προσέξουμε να μην έχουμε αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και ο κύριος Σμίτα θέλει να διασφαλίσει πλεονεκτήματα και για το μέλλον. Τέλος, πιστεύει ότι οι κανόνες μη προτιμησιακής ε, προέλευσης είναι σημαντικοί. Οι νομοθετικές προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν σαφείς κανόνες και ορισμούς με μια ισορροπημένη συμβιβαστική λύση με την ε, εισηγήτρια και του συναδέλφου ε, θα επιτευχθεί. Είναι βέβαιος γι' αυτό. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και να επιβεβαιώσω ότι η ομάδα μου συμφωνεί με τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Απλώς δεν προλάβαμε χρονικά για να υπογράψουμε, αλλά συμφωνούμε. Αυτό θέλω να το διευκρινίσω για να είναι σαφές ότι η μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου στηρίζει τις τροπολογίες σας στο λευκό κομμάτι. Αυτό θέλω να το διευκρινίσω σαφώς. Επίσης πιστεύω ότι οι τροπολογίες της εισηγήτριας είναι ισορροπημένες και δεν είναι απλό να γίνει αυτό γιατί είναι πολλά τα συμφέροντα που αντιπροσωπεύονται εδώ που είναι μεγάλα οικονομικά συμφέροντα βεβαίως και είναι και συμφέροντα ασφαλείας. Προσπάθησε η εισηγήτρια πραγματικά να υποβάλει μια ισορροπημένη έκθεση. Θέλω να υπησέλθω σε κάποια θέματα όπως και ο κύριος Σμιτ το ζήτημα του, των κανόνων καταγωγής ε, πρέπει να προσέξουμε πολύ ώστε σε νομικό επίπεδο η ρύθμιση να είναι απόλυτα ε, ξεκάθαρη γιατί αν δεν έχουμε ασφάλεια δικαίου τότε θα δημιουργήσουμε περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα λύσουμε. Έκλειση λοιπόν ε, σε σχέση με κάποιες τροπολογίες. Νομίζω ότι για τους κανόνες καταγωγής πρέπει να υπάρχουν πολύ ξεκάθαροι νομικοί ορισμοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μακλάρκιν. Εξ ονόματος της κυρίας Μπίλεν, πολύ σύντομα για τις προτινόμενες τροπολογίες, επειδή θα συνεργαστούμε με την εισηγήτρια και τους σκιώδεις για να επεξεργαστούμε το κείμενο και ελπίζουμε να έχουμε μια θέση στην Επιτροπή, όπως κάναμε όταν δουλέψαμε για την έκθεση εξυγχρονισμού των τελωνίων. Πολλές τροπολογίες κατατέθηκαν πάνω στο καθεστώς ΑΑ και ο κύριος Μπίλεν με συναδέλφους άλλους ε, όπως ε, αναφέρθηκε, θέλουμε ε, απλοποιήσεις στους, στις επιχειρήσεις που έχουν AEO, γιατί αυτές οι επιχειρήσεις είναι αξιόπιστες. Για τους κανόνες καταγωγής το λευκό κείμενο θα πρέπει να εξεταστούν, αλλά νομίζω ότι μια συμβιβαστική διατύπωση είναι θέμα συνεργασίας μεταξύ σκιωδών, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει και εδώ ε, Γενική Συμφωνία για το άρθρο 62 και τη μέθοδο της, ε, του πετρελονιακής αξίας, του προσδιορισμού της αξίας. Δεν ξέρω για την, ε, ποια είναι ακριβώς η θέση της εισηγήτριας. Εγώ είμαι υπέρ της προσέγγισης που δεν θα επηρεάσει αρνητικά την νοσιακή οικονομία. Τέλος, οι τροπολογίες <clears throat> που αφορούν εκτελεστικές και κατεξουσιοδότηση πράξεις ε, δεν θα αποφασίσουμε ακόμα πριν συζητήσουμε με την εισηγήτρια και τους σκιώδεις. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλα μέλη που θέλουν να μιλήσουν εκτός από τους σκιώδεις. Όχι. Εν τη αυτή περιπτώσει καλώ την Κομισιόν να μας πει αν θέλει κάτι και για το λευκό κείμενο, αν μπορείτε να επιβεβαιώσετε επίσημη συμφωνία με την Κομισιόν εδώ, σε αυτό το στάδιο, είναι λεπτά θέματα σε σχέση με την επίσημη συμφωνία. και εγώ συνάντησα την Κομισιόν για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Γίνεται ένα ενεργό διάλογο με την Κομισιόν και το Συμβούλιο και ελπίζω ότι θα επιτελεστεί πρόοδο. Ε, η Κομισιόν, λοιπόν, παρακαλώ να σχολιάσει την έκθεση και τα όσα άκουσε από τη συζήτηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι γνωρίζετε το χρονοδιάγραμμα για την εξέταση της πρότασης και για να ολοκληρωθεί είναι πραγματική πρόκληση για όλα τα θεσμικά όργανα και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας και εσάς κύριε Πρόεδρε και την ε, εισηγήτρια και όλα τα μέλη και τις προσπάθειες που κατέβαλαν ώστε να τηρήσουν αυτό το πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Ελπίζω ότι θα έχουμε τον ίδιο ενθουσιασμό από την άλλη πλευρά, δηλαδή από την νομοθετική πλευρά. Σχετικά με την παρουσίαση που έγινε από την εισηγήτρια και τα σχόλια των σκιωδών εισηγητών, το θέμα των λευκών και των γκρίζων τμήματων. Θα ήθελα να σας πω κύριε Πρόεδρε ότι εν πάση περιπτώσει στο παρόν στάδιο της διαδικασίας η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να τοποθετηθεί επίσημα ούτε επί των λευκών ή ούτε επί των γκρίζων τμήματων. Ε, μπορεί να συζητηθεί τι είναι το λευκό τμήμα. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Η συγγήτρια μας είπε ότι πολλές τροποποιήσεις που έγιναν όσον αφορά τις προσωρινές Κατά αναποθέσεις μπορεί να αφορούν τα λευκά τμήματα. Για την Επιτροπή αυτό δεν είναι σίγουρο, διότι η ίδια η Κομισιόν έκανε ε, μία ε, πρόταση τροποποιώντα τον εξοχρονισμένο τελωνιακό κώδικα. Συνεπώ αυτό είναι ένα τομέας όπου τα περιθώρια συζητήσεων και διαπραγματεύσεων είναι μεγάλα. Εν πάση περιπτώσει όμως, και το αναφέρατε κι εσείς, το γεγονός ότι ο νομοθέτης παρέμβει σε θέματα που δεν ήταν αντικείμενο της πρόταση επιτροπή Επιτροπής είναι ένα λεπτό θέμα το οποίο περιλαμβάνεται στη Διαθεσμική Συμφωνία και η Επιτροπή θα προτιμήσει να δει την θέση και αν είναι δυνατόν τη ενιαία συνενετική θέση των θεσμικών οργάνων για να δει σε ποιο βαθμό μπορεί να αποδεχθεί αυτές τις τροποποιήσεις. Ω προ την ουσία, πάλι δεν θέλω να επισέλθω στις ε, λεπτομέρειες των τροπολογιών, επειδή δεν είμαι εξειδοτημένο προ τούτο, αλλά σχετικά με ορισμένα σημεία γενικά, γενικής φύσης που ανέφεραν οι παρεμβαίνοντε, όσον αφορά την βελτίωση, την αναβάθμιση της θέσης ε, του οικονομικού φορέα, του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα. Βεβαίω, αυτό ε, υπάρχει. Το ζητούμενο εδώ είναι μάλλον κατά πόσον τα στοιχεία, οι προϋποθέσεις που έχουν σχέση με τη χορήγηση αυτού του καθεστώτος, ιδιώτες ή τα ωφέλη που απορρέουν από αυτό το καθεστώς θα πρέπει να καθυλωθούν, να προσδιοριστούν στη βασική πράξη ή κατά πόσο δεν θα πρέπει να έχουμε ορισμένα περιθώρια ελιγμών για να προσαρμόζονται στις καταστάσεις, στις ανάγκες όσον αφορά τους ελέγχους αλλά και την πρόσβαση σε ορισμένες άδειες. Από αυτή την άποψη δεν υπάρχει διαφορά προς την προσέγγιση μεταξύ των θεσμικών οργάνων, κοινοβουλίου δηλαδή και επιτροπής. Απλώς πρέπει να διατηρηθεί η ισορροπία, όπως είπε η συγγήτρια πολύ σωστά. Έρχομαι τώρα σε ένα θέμα που αναφέρθηκε επίσης. Για την Επιτροπή, για το Κοινοβούλιο, η ιδέα την οποία ε, συμμερίζονται και ορισμένα μέλη του Συμβουλίου να περάσουν ορισμένε διατάξει που μέχρι τότε ήταν εφαρμοστικέ διατάξει στο επίπεδο τη ε, βασική πράξη, να διατηρηθεί στην βασική πράξη διατάξει που βρίσκονται στον τελειακό κώδικα, στο σημερινό τελειακό κώδικα. Και αυτό είναι θέμα πώς μπορεί να σταθμίσει κανείς ε, τα υπέρ και τα κατά, να βρει τη σωστή ισορροπία. Η Επιτροπή πιστεύει ότι ναι, οπωσδήποτε γνωρίζουμε ότι ο νομοθέτης δεν είναι υποχρεωμένος να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή. Αλλά από την άλλη πλευρά, εάν οι διατάξει είναι αρκετά σταθερές, αρκετά γνωστές και δεν χρειάζεται να συζητηθούν και επιτρέπουν να δοθεί μεγαλύτερη νομική σαφήνεια και ασφάλεια στους χρήστες, είτε θεωρούνται ουσιαστικά ούτε όχι, αυτό δεν είναι το ζητούμενο, τότε αυτοί οι κανόνες μπορούν να διατηρηθούν ε, στην βασική πράξη. Πάντοτε διατηρώντας ε, την ισορροπία και την ευελιξία που απαιτείται προκειμένου ο κανονισμός να προσαρμοστεί στις διάφορες καταστάσεις και στην εξέλιξη του οικονομικού κλίματος. Για το θέμα της ευθυγράμμισης και της επιλογής των διαδικασιών, ε, δηλαδή επιτροπολογία ή όχι, αυτό είναι ένα τομέα ιδιαίτερα ευαίσθητο, όπω αντιλαμβάνεστε, εφόσον η ανάγνωση τη συνθήκη, η εφαρμογή τη συνθήκη, στην προκειμένη περίπτωση, κατά περίπτωση μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές αναλύσεις. Η Επιτροπή εδώ θα προτιμούσε να περιμένει, ούτω ώστε η Επιτροπή σα και το Κοινοβούλιο να σκεφτούν καλά το θέμα και να αποφασίσουν ποια θα είναι η μορφή εξοδότηση που θα δοθεί στην Επιτροπή για την α ή β διάταξη. Θα περιμένει να δει τι θα πει και το Συμβούλιο και ανάλογα με τις συγκλήσεις, με τις αποκλήσεις μεταξύ των δύο πυλώνων, θα δει ποια θα είναι η δική της τοποθέτηση και ενδεχομένως κατά πόσον αυτό το θέμα θα είναι σημαντικό για να συζητηθεί σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου. Τέλος, Πρόεδρε, θα, θα τελειώσω από εκεί που ξεκίνησα. Δηλαδή ότι οι εργασία σας προχωράνε πολύ καλά. Νομίζω ότι το χρονοδιάγραμμα ε, από το Κοινοβούλιο ακολουθείται σωστά. Αναμένουμε από το Συμβούλιο να προχωρήσει με ανάλογο ρυθμό και φυσικά η θέση της Επιτροπής και αυτό που ζητά ρητά η Επιτροπή όχι μόνο για ε, λόγω των νομικών προθεσμιών, δηλαδή ε, το τέλος του 2013, αλλά το γεγονός ότι οι χρήστες του τελωνιακού κώδικα πρέπει να γνωρίζουν ποιο θα είναι το νομικό πλαίσιο των δράσεών τους στο ταχύτερο δυνατόν. Η Επιτροπή λοιπόν συνηγορεί πάντοτε υπέρ της στήρησης ε, του αρχικού χρονοδιαγράμματος προκειμένου αυτός ο κώδικα να υιοθετηθεί όπως είχε προβλεφθεί για να αρχίσει να ισχύει πριν από τον Ιούνιο 2013. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση και τις διευκρινήσεις εκεί όπου υπάρχει ένα περιθώριο ελιγμών, για να το πω λεπτά, στις ε, λευκές περιοχές. Τώρα για τις κατεξουσιοδότηση και εκτελεστικές, μέχρι τώρα είναι μία κραγίσα βόμβα και η συγγήτρια θα πρέπει να εκτονώσει το θέμα αυτό για να μιλήσω με αυτή την ορολογία. Θα συνοψίσετε λοιπόν τώρα που βρισκόμαστε, θα απαντήσετε ίσως και στους συναδέλφους και στην Κομισιόν. Η συγγήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε, εντάχει. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που μίλησαν, τους χιόντις εισηγητές ή όσους ε, τους αντικατέστησαν. Τους ευχαριστώ όλους λοιπόν για τα επικοδομητικά τους σχόλια που αποδεικνύουν ότι το πνεύμα συνεργασίας και κοινή δουλειά, α πούμε, μας διέπει πάντοτε, διότι γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε απέναντι σε ένα περίπλοκο τεχνικό θέμα με χιλιάδες επιπτώσεις ε, σε πολλούς εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους και γι' αυτό το λόγο πρέπει να μετακινούμε άρθρα, τμήματα άρθρων με μεγάλη σύνεση, προσοχή, επειδή ο διάβολος κρύβεται τις λεπτομέρειες, όπως λέμε μερικές φορές. Και συνεπώς πρέπει να είμαστε επάγρυπνοι, προσεπτικοί και να παρακολουθούμε, να ακούμε πραγματικά τα μηνύματα των φορέων, αρχικά των οικονομικών φορέων και όλων των άλλων διαφερομένων, τον επιχειρηματικό κόσμο, μικρομεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις, εργαζόμενο κόσμο, ώστε να κάνουμε τις σωστές προσαρμογές, να βρεθούν οι σωστές ισορροπίες. Τα όσα υπόθηκαν σήμερα το πρωί αποδεικνύουν τον προβληματισμό μας και τη βούληση να προχωρήσουμε μαζί με τρόπο λογικό, συνειδητό και ισόρροπο. Τους ευχαριστώ όλους επίσης, όλους και όσες υποστήριξαν και επιβεβαίωσαν την υποστήριξή του σε ορισμένες τροπολογίες ουσίας που καταθέσαμε όσον αφορά την προσωρινή αναπόθεση, ε, την ε, αναβάθμιση του καθεστώτος ε, του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα. Υπάρχουν ορισμένα θέματα, το είπα, το ξαναείπαμε, επί των οποίων πρέπει να βρούμε τις σωστές προσαρμογές, την συμφωνία, τη σωστή συμφωνία, τον συγχρονισμό, όπως ε, η ηλεκτρονική υποστήριξη, τα ηλεκτρονικά μέσα για τις ταμιακές διοικήσεις, για την άρση μη των υποχρεώσεων, για την εγκατάσταση ε, στην επικράτεια της Ένωσης τους κανόνες ε, καταγωγής. Ε, ναι, υπάρχουν, ε, έχει γίνει εδώ πρόοδος, πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο και να επιδείξουμε μεγαλύτερη πνευματική δημιουργικότητα για να βρούμε σαφείς, συγκεκριμένους, χρήσιμους κανόνες που δεν θα δημιουργήσουν αστάθειες, ασάφειες και ανασφάλειες. Μεγάλο θέμα, το γνωρίζω. Άκουσα πολύ προσεκτικά τα μηνύματά σας, κυρίως τα μηνύματα της κυρία Ρούλερ και του κυρίου Σμιτ, του εκπροσώπου μάλλον του κυρίου Σμιτ. Θα σταματήσω εδώ, τελειώνοντας με το θέμα της συνέχισης των εργασιών μας για την κατανομή των αρμοδιοτήτων το λεπτό και ευαίσθητο θέμα μεταξύ βασικών κειμένων, πράξεων, κατεξιοδότηση, εκτελεστικών πράξεων. Γνωρίζω ότι πρέπει να σταθμίσουμε, να ισορροπήσουμε τη θέση μας και να δουλέψουμε ε, με γνώμονα ε, την νομική σαφήνεια και μπορούμε να διασφαλίσουμε, να καθησυχάσουμε τα άλλα θεσμικά όργανα ότι αυτό το πνεύμα μας διέπει. Άλλωστε δεν συμβαίνει αυτό μόνο στη δική μας Επιτροπή. Σίγουρα θέλουμε πάντοτε να ακολουθήσουμε μια γραμμή με βάση τη σύνεση. Αλλά τελικά πρέπει όχι μόνο να βρούμε μια ισορροπημένη λύση, αλλά να συντάξουμε ένα κείμενο το οποίο να μην είναι πολύ μεγάλο, υπερδιογκωμένο από τμήματα που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, πρέπει να επανεισαχθούν ουσιαστικέ διατάξει στο βασικό κείμενο, αλλά κατόπιν να γίνει η απαραίτητη προσαρμογή με τι δύο άλλες πράξει που είναι οι πράξει κατεξιοδότηση και εκτελεστικέ πράξει. Αυτέ οι δύο πράξει είναι πολύ πολύ σημαντικά στοιχεία επί των οποίων πρέπει να παίξουμε αν θέλετε με ευθεία προκειμένου να ενσωματώσουμε τα απαραίτητα στο βασικό κείμενο, κείμενο το οποίο θα πρέπει να είναι ευανάγνωστο, σαφές για εκείνους για τους οποίους προορίζεται, κυρίως ωραία οι τελωνιακές διοικήσεις, αλλά ο επιχειρηματικός κόσμος ο οποίος χρειάζεται σταθερότητα, σαφήνεια και απλούστευση. Θα σταματήσω εδώ. Όπως σας είπα, αντιμετωπίζουμε την πρόκληση να πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μας και θα προτείνουμε πολύ σύντομα μία ημερομηνία συνεδρίασης των σκιωδών εισηγητών κατά ε, την Ολομέλεια του Στρασβούργου και γνωρίζουμε ποιο είναι το δικό μας χρονοδιάγραμμα, δηλαδή η ψηφοφορία της έκθεσης και ελπίζουμε θα τηρηθεί αυτή η προθεσμία και θα κάνουμε τα πάντα για να τηρήσουμε τις προθεσμίες μας. Προβλέπετε λοιπόν αυτή η ημερομηνία για τις 18 Δεκεμβρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Good. Ευχαριστούμε πολύ. Στις 17 ε, θα γίνει μια σημαντική προκαταρκτική συζήτηση. Θα συζητήσουμε με τους ε, συγητές και το Συμβούλιο για να υπάρξει συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Εξαρτάται από τους συζητητές και τις πολιτικές ομάδες βέβαια και εν ώψη της σημασίας αυτού του θέματος αλλά και του χρονοδιαγράμματος αν αποφασίσετε με τους εισηγητές θα παρουσιάσετε μία πρόταση που μπορεί ταυτόχρονα να εγκριθεί. Το λέω αυτό δημοσία στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος, γιατί καμιά φορά οι διαδικασίες για τη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση δεν είναι τόσο ε, ξεκάθαροι, ενώ εμείς ε, τα είπαμε όλα πολύ ε, συγκεκριμένα και το χρονοδιάγραμμα το προβλέπει αυτό ως δυνατότητα. Εξαρτάται από εσά και τους κοιόδης και η προσέγγιση, η προσέγγιση σας ως προς και κατεξουσιοδότηση πράξης είναι καλές. Θα καλέσουμε την Γραμματεία να συνεργαστεί μαζί σας και να είναι απόλυτα σαφές ότι οι πράξεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν για το σωστό σκοπό. Γιατί αυτή είναι η συζήτηση που διεξάγεται τώρα και όπως ξέρετε τώρα η Κομισιόν πήγε το Κοινοβούλιο στο δικαστήριο και υπάρχει τώρα μια υπόθεση που εξελίσσεται σε σχέση με αυτό που θεωρεί η Κομισιόν ε, κακή κατανομή των εκτελεστικών και κατεξουσιοδότηση πράξεων. Περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Δεν αστειευόμουν όταν είπα ότι αυτή είναι μια, μια κραγίσα βόμβα, γιατί μπορεί το Κοινοβούλιο να παίξει το ρόλο του καταλήτη για κάποια θέματα εδώ. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να συμφωνήσουμε σε μια, στην εφαρμογή όλων αυτών των θεμάτων. Η γραμματεία μου θυμίζει ότι όλοι έχουν αντίγραφο των του κανονισμού από τον Ιούλιο του 2010 που περιέχει σαφείς κανονισμούς. Καλό είναι να τα δούμε αυτά, γιατί καμιά φορά συζητάμε σαν να είναι όλα αυτά αφηρημένα θέματα. Μέρος του προβλήματος τώρα πιστεύω ότι είναι ότι τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι η κατεξουσιοδότηση πράξεις δεν είναι αρκετά ανοιχτές ώστε να συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις Και υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ε, που είναι αφέρεται σε σχέση με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις, τις συμφωνίες ε, που πρέπει να επιτευχθούν. Τώρα η Κομισιόν επιδιώκει οριζόντια συμφωνία με Συμβούλιο και Κοινοβούλιο για τις πράξεις αυτές για να λυθεί το πρόβλημα. Πρέπει να πω ότι εν ώψη της σημασίας του θέματος νομίζω ότι δεν προχωρούμε όπως πρέπει. Έτσι λοιπόν λάβετε το υπόψη εσείς που συνεργάζεστε με την Προεδρία. Στο ενδιάμεσο σας ευχόμεθα σε εσά και στην ομάδα που θα ασχοληθεί με το θέμα καλή επιτυχία στις επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες για να λυθεί το θέμα. Μπορεί να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή της συζήτησης για τις εκτελεστικές και τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξης. Βάλτε, ε, πάρτε προστατευτικά μέτρα, ε, βάλτε ε, στο κεφάλι σας προστατευτικό κράνος ε, για να αποφύγετε τα χτυπήματα. Ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε στο επόμενο θέμα που είναι ο ενεργειακός, οδικός, ο ενεργειακός χάρτης πορείας. Ο κύριος Σμιτ είναι μακριά με την αντιπροσωπεία των χωρών ΑΚΕ, αλλά ο κύριος Χατζημαρκάκης είναι πάντοτε παρόν και εκείνος θα μας μιλήσει εξ ονόματός του. Να καλωσορίσω και τον κύριο Γουέστροπ, νομίζω, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ο αρμόδιος εδώ, λοιπόν, από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας για να απαντήσει σε πιθανές ερωτήσεις αργότερα. Να δω και ποιος είναι εδώ από του κοιόδη ηγητέ. Ο καθηγητής Κορέια Ντεκάμπος ε, είναι εδώ. Η κυρία Μπάστος είναι εδώ. Η κυρία Ρούντερ. Η κυρία Μακλάρκιν. Εκτός αν και μας δώσει και τις σημειώσεις της φεύγοντας, ο κύριος Μπίλαν, ο κύριος Χατσμαρκάκης καταρχάς για να ξεκινήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος του κυρίου Σμιτ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και όδης για την ε, αγαστή συνεργασία, όπως ξέρετε θα ψηφίσουμε αυτό το σχέδιο κειμένου ε, σήμερα το απόγευμα. Υπάρχουν κάποια σημεία βέβαια ε, στα οποία τα, κράτη, τα μέλη δεν μπορούν να συμφωνήσουν και ένα από αυτά είναι η φύγης ενέργεια και ο συντάκτης ε, θεωρεί ότι η πυρηνική ενέργεια θα είναι σημαντική και για το μέλλον μη συμβατικέ ε, τεχνολογίε, όπω για παράδειγμα η δέσμευση και η αποθήκευση του άνθρακα, είναι σημαντικέ και θα απασχολήσουν το κοινό στο μέλλον. Θα πρέπει όμω να αφήσουμε και νομοθετικό περιθώριο για μελλοντικέ γνώσει και τεχνολογία και όλοι Σμιτ πιστεύει ότι θα καταφέρουμε να επιτύχουμε μια ισορροπημένη συμβαστική πρόταση. Θα πρέπει να είναι ε, τα πάντα κατάλληλα για την ενέργεια για του καταναλωτέ και για τι επιχειρήσει. Ε, ενδιαφέρουν οι ενεργειακοί φόρου, και η ανταλλαγή εκπομπών είναι βασικός στόχος για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να μην πιέζονται οι πιο ευάλωτοι ε, καταναλωτές. Τα εφή δίκτυα είναι το μέλλον. Η ε, παιδεία και η ενημέρωση των καταναλωτών είναι σημαντικές και θα πρέπει να διατίθεται πληροφορίες και για τους καταναλωτές και για τους επιχειρηματίες. Επίσης, ε, θέλουμε να έχουμε καλή ενεργειακή απόδοση και για την ε, ε, αποτελεσματικότητα της ενέργειας και ε, για τις μελλοντικές μας προτάσεις. Θέλουμε να βοηθήσουμε την εσωτερική αγορά ενέργειας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Να ακούσουμε τους και οδησίτης. Ο καθηγητής Κορέα Δεκάμπος θα λάβει πρώτος το λόγο. Υπάρχουν πάρα πολλές αλληλοεπικαλύψεις στις συνεδριάσεις των Επιτροπών σήμερα και λείπουν αρκετοί. Ο κύριος Κάμπος. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που μου επέτρεψαν να ξεκινήσω. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Όλε Σμιτ για την πολύ καλή δουλειά που κάνει ε, σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Είναι αρκετά σημαντικό το έγγραφο αυτό, διότι θα διαμορφώσει το μέλλον για τα επόμενα 35 χρόνια και είναι πάρα πολύ σημαντικό και από στρατηγική σκοπιάς. Η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών υποστηρίζει ε, αρκετές τροπολογίες, διότι είναι επεπισμένη ότι θα προσφέρουν σαφήνεια στο κείμενο. Δυστυχώς ε, δεν θα μπορέσω να συμμετέχω στην ψηφοφορία σήμερα το απόγευμα, αλλά... Ε, επιθυμώ να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα διότι η θετική έκβαση θα μας βοηθήσει να έχουμε μια εσωτερική αγορά ενέργειας με κοινούς κανόνες, διαφάνεια, ανταγωνισμό, ε, εναρμόνιση, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο της ασφάλειας εφοδιασμού, βιωσιμότητας του περιβάλλοντος και ευρύτερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσω της καλής λειτουργίας των Εθνικών Ρυθμιστικών Φορέων και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού. Ο βασικός στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι οι τιμές για τους καταναλωτές θα μειωθούν και βεβαίως γνωρίζουμε ότι μέσω αυτής της έκθεσης χρειάζεται να γίνουν και αρκετές αλλαγές, διότι είναι πολύ παλιό το δίκτυο και χρειάζεται ανανέωση. Ελπίζουμε όμως στο εγγύς μέλλον οι τιμέ για τους καταναλωτές να μειωθούν. Να σας πω και κάποια καλά νέα. Εχθές ε, αργά το απόγευμα καταλήξαμε σε συμφωνία στις στον τριμερή διάλογο για τα δίκτυα ενέργειας. Η συμφωνία αυτή ε, είναι ακόμα ένα ανεμονή της τελικής έγκρισης και του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βεβαίως. Και το Σώμα των Επιτρόπων θα πρέπει να την εγκρίνει, αλλά ε, παρόλα αυτά καταλήξαμε σε μια τεχνική συμφωνία και η συμφωνία αυτή είναι υπέρ της ε, ανάπτυξης μιας εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Και εδώ να πω ότι τα βασικά προσκόμματα προς την εσωτερική αγορά, το λέω αυτό με πάσα προσοχή, ε, αλλά να σας πω ότι εγώ δεν είμαι με το μέρος του Κοινοβουλίου τουλάχιστον για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, δεν χρειάζεται να κωδικοποιήσετε το μήνυμά σας, σας καταλάβαμε. Η κυρία Μπάστος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω πορτογαλικά, διότι υπάρχει διερμηνία. Πολύ σοφή απόφαση να υπάρχει διερμηνία λέει ο Μιλήτρια. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον συνάδελφο Όλε Σμιτ, παρά το γεγονό ότι δεν μπορεί να είναι παρόν εδώ σήμερα, γιατί ε, μας παρουσίασε ε, πάρα πολύ καλέ συμβιβαστικέ προτάσει. Να ευχαριστήσω και του υπόλοιπου και όδης ε, διότι ήταν διατεθειμένοι να... Ε, ε, συμβιβαστούν και είχαμε ένα διάλογο ο οποίος πραγματικά συνεισέφερε στο έργο μας. έχουμε έξι λοιπόν συμβιβαστικές τροπολογίες για έξι σημεία τα οποία αποτελούν κλειδί για τη συγκεκριμένη έκθεση, για τα θέματα ανταγωνισμού, την ενεργειακή αυτάρκεια, το, ε, τις επιπτώσεις του άνθρακα, τα δίκτυα ε, των καταναλωτών και το θέμα του ενεργειακού εφοδιασμού και των τιμών της ενέργειας. Οι τροπολογίες αυτές είναι οι τροπολογίε τι οποίε καταλήξαμε κατόπιν συνένεση και ε, ε, επιμείναμε ιδιαίτερα στη διατύπωση. Φαντάζομαι λοιπόν ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα στην ψηφοφορία σήμερα το απόγευμα. Ω ε, σκιώδη συγγήτρια του ΕΛΚ ζητώ ε, να ψηφίσουμε την τροπολογία 24 στην οποία ζητούμε να μην υπάρχει κατακαιρματισμό όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών ε, από τα βιοκαύσιμα και εκεί ζητούμε τη διαγραφή του όρου εθνικός. Επομένως, ζητήσουμε κατά τμήματα ψηφοφορία και επίσης υπάρχει και όρος δημόσιο στην τροπολογία 26, τον οποίο ζητήσαμε διότι δεν θέλαμε να είναι τόσο κλειστή και περιορισμένη και το ΕΛΚ έχει ε, παρουσιάσει μια ρεαλιστική αντιπρόταση ώστε να μην αποκλειστεί καμία ενεργειακή πηγή από το ενεργειακό μας μείγμα. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι το ΕΛΚ ήταν διατεθειμένο να καταλήξει σε συνένεση, γεγονός που ήταν καθοριστική σημασίας. διότι ε, αποσύρθηκε η τροπολογία 18, η οποία διευκόλυνε στη συνέχεια τις διαπραγματεύσεις και μπορέσαμε να έχουμε συνένεση για όλες τις υπόλοιπες ε, συμβαστικές τροπολογίες. Η τροπολογία 36 ήταν καθοριστική σημασία ώστε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό τον οποίο προσυπογράφω και εγώ και, ήταν, και πρόκειται για τη συμβιβαστική πρόταση υπεριθμών 6. Να ευχαριστήσω λοιπόν και πάλι τον συνάδελφο Όλε Σμιτ και όλους όσους ε, συνεργάστηκαν για τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση και ελπίζουμε η Επιτροπή Ήτρε να συμπεριλάβει τις προτάσεις μας στην έκθεσή της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρούλε. Θα είμαι σύντομη. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σμιτ για τις πολλές προτάσεις για την έκθεση, για τις συμβιβαστικές προτάσεις. Εμείς ως ομάδα όμως δεν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με την τροπολογία αυτή, γιατί το θέμα το πυρηνικό είναι καθοριστικό για μας και νομίζω ότι εν ώψη των μεγάλων οικονομικών αναγκών που έχουμε στην αποθήκευση και στα δίκτυα, θα πρέπει να κάνουμε εκεί τις επενδύσεις και όχι σε ε, πεδία όπως πυρηνική ενέργεια ή δέσμευση, αποθήκευση ε, άνθρακα, ε, του άνθρακα και γι' αυτό δεν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Κατανοούμε τη θέση σας. Ε, ένα σημείωμα ε, για τον κύριο, τον κύριο Μπίλαν και θα την αναφέρω σε λίγο. Θα την αναφέρω. Ο κύριος Μπίλαν λέει ότι είναι πολύ ικανοποιημένο από το κείμενο και τις συμβιβαστικές τροπολογίες και θα ψηφίσει υπέρ γιατί θεωρεί ότι είναι πολύ ισορροπημένο το κείμενο. Οπότε θα υποστηρίξει ε, τον εισηγητή και την συμβιβαστική δύο που τονίζει την εσωτερική ενεργειακή αγορά και αναφέρει την ανάγκη μείωση εξάρτηση από τρίτες χώρες και επίσης ε, ε, στην συμβιβαστική τροπολογία 5 και αν και δεν αναφέρονται μη συμβατικές πηγές ενέργειας, παρόλα αυτά θα στηρίξουμε τον εισηγητή. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που θα ε, προωθήσουμε το κείμενο. Και τώρα ο κύριος Χάντλ, ο τελευταίος σκιώδης, κύριε Χάντλ, δεν θα μιλήσετε θα μιλήσετε. Ήθελα να σας καλωσορίσω και στην Επιτροπή ως καινούριο μέλος από την ομάδα σας, γιατί νομίζω ότι πρώτη φορά έρχεστε. Λοιπόν, άλλος κανείς θέλει να συμβάλλει στη συζήτηση. Όχι. Ο κύριος Βέστροπ από την Κομισιόν θα μιλήσει και μετά ο κύριος Χατζημαρκάκης θα συνοψίσει εξ ονόματος του κυρίου Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σχετικά σύντομος. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις συζητήσεις που έγιναν στην Επιτροπή σας για αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Το σχέδιο γνωμοδότησης από τον εισηγητή ευθυγραμμίζεται και με τις σκέψεις της Κομισιόν ιδιαίτερα τη σημασία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας που αναφέρθηκε και σήμερα. Είναι πολύ κεντρικό το θέμα για μας. Ξέρετε ότι η Κομισιόν έκανε πριν από λίγες εβδομάδες ανακοίνωση για το θέμα όπου αναγνωρίζουμε 100% τη σημασία της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς όχι μόνο για αυτό το θέμα, αλλά για να αποτελέσει τη βάση ενεργειακή αγορά για να πετύχουμε τους άλλους στόχους της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, ανταγωνιστικότητα, ασφάλεια εφοδιασμού κλπ. Σημειώνω τις συζητήσεις ε, για, τα θέματα που θέσατε για το CCS και την πυρηνική ενέργεια. Δεν μας εκπλήσει ότι δυσκολεύεστε να συμφωνήσετε ε, εδώ. Λοιπόν, μετά από αυτά νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε μπορεί να συνεχιστεί, να γίνει ψηφοφορία σήμερα το απόγευμα. Ο κύριος Μαρκάκης. Όπως είδαμε και ακούσαμε και από τις συζητήσεις, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ισορροπία σε αυτό το στρατηγικό και δύσκολο τομέα. Όλες Σμιτ όμως νομίζω ότι κατάφερε να κρατήσει μια ισορροπία, παρόλο που καταλαβαίνω ότι βέβαια η ομάδα των Πρασίνων δεν θα μπορέσει να ψηφίσει υπέρ. Ε, να σας ευχαριστήσω όλους και να υπογραμμίσω ότι η ολοκλήρωση της ενεργειακής εσωτερικής αγοράς ε, όχι μόνο σε αυτός ο σκοπός, ε, έχει τεράστια σημασία και η Επιτροπή ΙΜΚΟ μαζί με την Ήτρε πρέπει να δουλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Επιβεβαιώνω ότι θα ψηφίσουμε στις 4 ε, σήμερα το απόγευμα έχει ετοιμαστεί ο κατάλογος, έχετε δει τις συμβιβαστικές. Θα σας δω λοιπόν το απόγευμα και τον κύριο Χατζημαρκάκη για να το ψηφίσουμε αυτό. Είναι γνωμοδότηση για την Επιτροπή Βιομηχανίας που είναι καθηλήν αρμόδια. Προχωρούμε. Το επόμενο θέμα μας είναι η γνωμοδότηση από την Επιτροπή για την απόσπαση των εργαζομένων. Έχουμε γλιτώσει πέντε λεπτά μέχρι τώρα, οπότε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Α, θα είναι σε ένα λεπτό. Η κυρία Τουρούνεν θα είναι εδώ σύντομα, οπότε θα αρχίσουμε. Μόλις έρθει, ελπίζω να έρθουν και οι συγητές, οι σκιώδεις συγητές. Ένα μικρούλι, μικρό διάλειμμα. Ε, κύριε Κοφράτη, εσείς θα εκπροσωπήσετε την κυρία Γκέπχαρτ, εντάξει. Uh, okay, ladies and gentlemen, I think, um... Ωραία, λοιπόν. I say I warmly welcome uh, Mrs. Turinen. Καλωσορίζω θερμά λοιπόν την κυρία Τούρινεν στην ε, συνεδρίασή μας. Είναι η συγγήτρια για τη γνωμοδότηση για την εφαρμογή της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων, ε, η οποία ε, απευθύνεται φυσικά στην Επιτροπή Απασχόλησης. Η συγκεκριμένη γνωμοδότηση έτυχε ιδιαίτερη προσοχή από τους συναδέλφους. Έχουμε 330 τροπολογίες ε, για τη γνωμοδότηση, κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθε σε γνωμοδοτήσει, οπότε καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι περίπλοκο και ενδιαφέρει πολλού. Ε, θα δώσω λοιπόν το λόγο στην Έμιλη Τούρινεν για να μας δώσει την άποψή της για τις τροπολογίες και ε, κατόπιν περιμένουμε και το σκιώδη συγκητή του ΕΛΚ, ο οποίος ε, φαντάζομαι ότι θα μας δώσει κάποιες εξηγήσεις, διότι το ΕΛΚ κατέθεσε πολλές από αυτές τις τροπολογίες και ελπίζω λοιπόν να είναι ο σκιώδης του συγκητής εδώ εγκαίρος για να συζητήσουμε. Ο κύριος Κοφεράτη θα μιλήσει εκ μέρους της κυρίας Γκέπχαρτ εγώ θα μιλήσω εκ μέρους ε, της δικής μας της ομάδος και δεν ξέρω αν ε, θα μιλήσει και κάποιος εξ ονόματος της ΓΚΟΕ, δεν ξέρω κύριος Χάνπορ. Να ζητήσω λοιπόν από την Έμιλη Τούρινε να, συνεχίσει τη συζή... να ξεκινήσει τη συζήτηση, να καλωσορίσω και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει κάποιος εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, την περιμένουμε ακόμα την Επιτροπή. Εντάξει. Αν υπάρξει λοιπόν εκπρόσωπος, θα είχαμε πει να ξεκινήσουμε στις 10 και 20. Ξεκινήσαμε στην ώρα μας σήμερα και ελπίζω να στείλει κάποιον εκπρόσωπο εν ευθέτω χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν τω μεταξύ όμως να ακούσουμε την κυρία Τουρνέν. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που ξεκινήσετε γέρος. Το εκτιμώ ιδιαίτερα, διότι πάντα είναι καλό να είμαστε ακριβείς. Έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες. Και όντως υπάρχουν επίμαχα ζητήματα στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά είμαι αισιόδοξη. Θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία και θα προσπαθήσω λίγο να σας ε, μιλήσω για τα διάφορα άρθρα εντάχει. Δεν θα μακρηγορήσω, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να σας δώσω κάποιες ε, πληροφορίες ε, ε, επί της ουσίας για το που θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες συμβαστικές προτάσεις. Για το άρθρο 1 που είναι η βασική ουσία, έχουμε κάποιες ε, τροπολογίες που αφορούν την εφαρμογή, ε, κάποιες τροπολογίες αναφέρονται στο δικαίωμα να παρέχει κάποιες υπηρεσίες ελεύθερα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε ότι στην ουσία πρόκειται και για τα δύο ζητήματα. Το θέμα είναι πόση έμφαση θα δώσουμε στο κάθε τμήμα και θεωρώ ότι εκφύσεως αλλά και λόγω του τίτλου είναι μια οδηγία για την εφαρμογή της απόσπασης των εργαζομένων, της οδηγίας από το 96. Επομένως, θέλουμε και να διασφαλίσουμε την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, αλλά και να υπάρχει κατάλληλη προστασία των εργαζομένων. Θεωρώ λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμβιβασμό σε αυτό το θέμα. Στο άρθρο 2 έχουμε τους ορισμούς. Και πάλι Θεωρώ ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία ώστε να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε όλα τα μοντέλα αγοράς εργασίας και το σκανδιναβικό μοντέλο και το γερμανικό και το μαλτέζικο. Θεωρώ ότι θα πρέπει να μιλάμε για αρμόδια αρχή φορέα, competent authority or body. Πρόκειται για κάτι το οποίο ε, συζητά και το Συμβούλιο, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε όλους ε, ο, τους παράγοντες που είναι απαραίτητοι για να καλέψουμε το συγκεκριμένο τομέα. Για το άρθρο 3, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αν ε, πρέπει κάποιος να πει ποιο είναι το πιο σημαντικό άρθρο, νομίζω ότι το άρθρο 3 είναι το πιο σημαντικό, το 12, το 9 και το 6. Δεν ξέρω αν ε, έχει γίνει εκ να το έχουμε και κατά καλή αριθμητική σειρά 3, 6, 9, 12. Τέλος πάντων, στο άρθρο 3 καθορίζεται πότε έχουμε απόσπαση εργαζομένου και πότε υπάρχει δυνατότητα διαφορετικής ε, ε, ε, κατάστασης και μπορεί να υπάρχει κατάχρηση στην κατάσταση αυτή. Υπάρχουν τροπολογίες εδώ προς διάφορες κατευθύνσεις για την ε, επιχείρηση απόσπασης υπάρχει ένας υποχρεωτικός κατάλογος και ένας ενδεικτικός κατάλογος, τον οποίο είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ ε, προτιμούσα να έχουμε έναν υποχρεωτικό κατάλογο, δηλαδή να υπάρχει ένας καθορισμένος ορισμός και από εκεί και πέρα να υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν προτείνει κάτι αντίστοιχο. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε κάτι ενδιάμεσο ίσως έναν υποχρεωτικό κατάλογο ο οποίος δεν θα είναι πλήρης, ώστε να υπάρχει και κάποιο περιθώριο για τα κράτη-μέλη ε, για την ε, de facto αξιολόγηση. Στο δεύτερο τμήμα τώρα για να αξιολογήσουμε κατά πόσον είναι όντως αποσπασμένοι οι εργαζόμενοι, ε, θα μπορούσαμε να έχουμε και πάλι ως συμβιβασμό έναν ε, αντίστοιχο κατάλογο. Προτάθηκε να έχουμε και ένα κλειστό κατάλογο, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο επικίνδυνο αυτό. Ο νομικός επιρρογνώμονας μας ε, έκρουσε τον κώδικα της προσοχής, διότι αν είναι πολύ ε, κλειστός ο ορισμός, δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε τι ισχύει στην πράξη και μπορεί να είναι επικίνδυνο αυτό. Καλό θα ήταν λοιπόν να έχουμε ένα κατάλογο ο οποίος δεν είναι πλήρης. Κατόπιν Τόσο εγώ όσο και άλλες πολιτικές ομάδες έχουν προτείνει την εισαγωγή ενός νέου άρθρου 3α που εξηγεί τι συμβαίνει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Θα ήθελα λοιπόν να προσθεθεί αυτό το άρθρο. Δεν ξέρω ε, αν οι άλλες πολιτικές ομάδες που δεν έχουν καταθέσει κάτι αντίθετο θα μπορούσαν να το ε, υποστηρίξουν, αλλά αυτό θα πρέπει να το δούμε στη συνεδριάση με τους Κιώδης για να δούμε αν μπορούμε να έχουμε ένα ε, νέο επιπλέον άρθρο. Για το άρθρο 4 δεν υπάρχουν τροπολογίες, δεν υπάρχουν λοιπόν και ανάγκη για συμβιβαστικές προτάσεις, είναι απλά τα πράγματα. Άρθρο 5. Και πάλι και εκεί δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Άρθρο 6, που είναι και πάλι σημαντικό άρθρο, έχουμε το χρόνο απόκρισης πότε θα πρέπει να απαντήσει ένα κράτος μέλος σε αίτημα άλλου κράτους μέλους, ποιο είναι το κατάλληλο χρονικό διάστημα και εκεί η κυρία Γκέπχαρτ πρότεινε να κατονομάζουμε τα κράτη-μέλη τα οποία δεν συνεργάζονται και δεν τηρούν την οδηγία. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα, αλλά όσον αφορά τα συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για κάτι πρακτικό. Μπορεί να υπάρχει κάτι επίγον. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 24 ώρες. Κάποιοι άλλοι έχουν προτείνει 2 ή 3 εργάσιμες. Θα πρέπει λοιπόν να είναι μια σύντομη λύση αλλά και πρακτική. Ε, δεν είναι καθόλου ιδεολογικής φύσεως, είναι κάτι πρακτικό το οποίο θεωρώ ότι μπορούμε να επιλύσουμε, αλλά καλό θα ήταν να υπάρχουν σαφείς προθεσμίες και νομίζω ότι το Συμβούλιο δεν θέλει να υπάρχουν προθεσμίες, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα έχουν προθεσμίες και οι διοικήσεις τους, αλλά κατ' εμέ είναι σημαντικό. Το άρθρο 7 επίσης ε, δεν έχει και σοβαρά προβλήματα. Και ε, περνάμε στο άρθρο 9 για τα εθνικά μέτρα ελέγχου. Η όλη συζήτηση και πάλι αφορά έναν κλειστό ή έναν ε, ανοιχτό κατάλογο. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι προτιμούν να έχουμε ένα κατάλογο ο οποίος δεν θα είναι εξαντλητικός. Ε, θα προσπαθήσω να μιλήσω με όλους για να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο να ε, βρίσκει σύμφωνο στους πάντες, ώστε να έχουμε ένα σαφή κατάλογο που να μπορούν να εφαρμόσουν επιχειρήσεις και να ξέρουν τι αναμένουν, αλλά από εκεί και πέρα και τα κράτη-μέλη να έχουν την ευελιξία να εφαρμόσουν διάφορες διαφορές ε, ίσως ας πούμε υποχρέωση να εκδίδονται, να δημοσιοποιούνται τα εθνικά μέτρα ελέγχου. Ε, είναι υποχρεωτικά κάποια πράγματα για, τα, για τις επιχειρήσεις, αλλά τα κράτη-μέλη έχουν ένα περιθώριο λιγμών. Ε, για το άρθρο 11 και 10... Άρθρα 10 και 11 δεν φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα. Το άρθρο 12 είναι ίσως το πιο δύσκολο άρθρο διότι αφορά την κοινή ε, και μερισμένη ευθύνη και δεν υπάρχει συμφωνία για το κατά πόσον θα πρέπει να παραμείνει, να διαγραφεί ή και να επεκταθεί, όπως πρότεινα εγώ στη γνωμοδότησή μου. Και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να γίνουν και περαιτέρω συζητήσει με τους κοιόδησίτες. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά προβλήματα σε γενικές γραμμές. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το άρθρο. Ίσως αποτελεί ε, εργαλείο. Θα μπορούσαμε ίσως να βρούμε και μια λύση δέουσας επιμέλειας. Για τα άρθρα 13, τώρα 14 και ούτω καθεξής δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Στο άρθρο 18... Ε, τις διμερείς συμφωνίες και ε, το σύστημα ε, μηχανοργάνωσης της εσωτερικής αγοράς, το IMI, ε, νομίζω ότι εδώ θα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στην πράση. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε τη χρήση του IMI, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει ε, μία ρήτρα sunset ε, για την εφαρμογή αυτού του συστήματος πληροφορικής υποχρεωτικά. Ε, αρκετές χώρες ε, θεωρούν ότι μπορούν να το χρησιμοποιούν ως συμπληρωματικό και εγώ δεν έχω πρόβλημα να χρησιμοποιηθεί έτσι. Καλό είναι να έχουμε ένα ισχυρό IMI. Ε, το οποίο θα μας βοηθήσει, αλλά να φτάσουμε μέχρι το σημείο να αποκλείονται οι διμερείς ε, ε συμφωνίες ε, νομίζω ότι είναι λίγο ακραίο. Ε, αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές όπως σας είπα νομίζω ότι το άρθρο 12 θα είναι το πιο ακαθόδες. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία στο τέλος, ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, θα μπορούσαμε ίσως να ε, το αφήσουμε στην Επιτροπή Απασχόλησης. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς μια απόπειρα ε, και κατά τα λοιπά είμαι αισιόδοξη. Well, thank you very much for... Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σαφέστατη επεξήγηση για το πού βρισκόμαστε με τις τροπολογίες. Είστε πολύ αποτελεσματικοί η γιατί συγκεντρώσατε του συναδέλφους για να βρεθεί συμβιβαστική λύση. Ιδιαίτερα στο άρθρο 12 πρέπει να ψηφίσουμε, γιατί ίσως υπάρχουν απόψεις που δεν γεφυρώνονται. Δεν πρέπει να μας φοβίζει η ψηφοφορία. Αυτό κάνει το Κοινοβούλιο. Άλλωστε εδώ υπάρχουν ε, ήδη κατατεθειμένες ε, ομαδικές ε, τροπολογίες μεταξύ πολιτικών ομάδων δηλαδή, που δείχνει ότι έχουν γίνει πολλές συζητήσεις. Η κυρία Τούν Σκιώδης θα μιλήσει για την κυρία Χάνσλη, ο κύριος Κοφεράτη, ο κύριος Τζόι. Εγώ θα μιλήσω για την ομάδα μου και έχω εδώ και από την κυρία Στράιτσεκ ένα γραπτό σημείωμα και τον κύριο Χάντλ. Η κυρία Τούν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πάρα πολύ διεξοδική δουλειά από την κυρία Τούρνεν. Ο κύριος Χαν, η κυρία Χάντσλικ έχει διαφορετικές πολλές απόψεις ε, σε σχέση με την κυρία Τούρνεν και τις, ε, μου τις έδωσε γραπτά. Θα τα διαβάσω λοιπόν στα πολωνικά. Η κυρία Χάντσλικ δεν είναι παρούσα σήμερα είναι στην ε, αντιπροσωπεία, με την αντιπροσωπεία στο ταξίδι στις χώρες ΑΚΕ. Θα διαβάσω λοιπόν αυτά που ετοίμασε. Η κυρία Χάνσλικ υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ ελεύθερης διακίνησης στην παροχή υπηρεσιών και την απόσπαση των εργαζομένων. Όλα τα μέτρα στην οδηγία πρέπει να είναι αναλογικά, όχι διακριτικά και καλά τεκμηριωμένα, αιτιολογημένα δεν πρέπει να δημιουργούν διοικητικό φόρτο. Η οδηγία για την εφαρμογή δεν θα πρέπει να εμπίπτει στην 96-71 ε, οδηγία ούτε να επηρεάσει την νομική βάση αρνητικά. Για την απόσπαση η κυρία Χάνσλικ πιστεύει ότι θα πρέπει να δούμε τις ε, αρμόδιες αρχές και να δούμε αν ο αποσπασμένος εργαζόμενος μπορεί να περιγραφεί ως τέτοιος. Δεν πρέπει να υπάρχουν αμφιβολίες και αυτό πρέπει να ισχύει για κάθε εργαζόμενο και κάθε επιχείρηση ώστε να προωθήσουμε την κινητικότητα της απόσπασης. Αυτό είναι σημαντικό για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά όμως δεν είναι υποχρεωτικά θέματα δεν ε, θα πρέπει να πληρούνται κάθε κριτήριο σε κάθε περίπτωση. Στο άρθρο 3, αυτά πρέπει να είναι ενδεικτικά στοιχεία, στοιχεία ανατολισμού και θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Για τα μέτρα ελέγχου τώρα όλα όσα αφορούν τον έλεγχο. Εδώ η κυρία Χάνσλικ πιστεύει ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα την ασφάλεια δικαίου αν έχουμε κλειστό κατάλογο μέτρων ελέγχου, θα πρέπει να δούμε πόσο αποτελεσματικά θα εφαρμόζονται στους διάφορους κλάδους αυτά τα μέτρα ελέγχου. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κατά την αξιολόγηση του κινδύνου. Ε, αυτή είναι η τροπολογία 159. Η κυρία Χάνσλικ πιστεύει ότι τα μέτρα ελέγχου και ο έλεγχος πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικά. Και επίσης θα είναι η έλεγχη αποτελεσματικότερη αν μετά τη σύναψη, μετά τον έλεγχο, την ολοκλήρωση του ελέγχου, η αρμοδιαρχή θα καταρτίζει ένα σημείωμα, ε, ούτως ώστε να υπάρχει προστασία των δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων και τις υποχρεώσεις. Ε, τώρα, περιγραφή των ισότιμων σχέσεων. Από την οδηγία 96-67. Ε, η εφαρμοστική οδηγία δεν μπορεί να αναφερθεί εδώ, γιατί πρόκειται για το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. 96-71 είναι η οδηγία. Ε, ό,τι αναφέρεται στην οδηγία αυτή πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένο. Στο σημείο 22 ε, του προημίου της πρώτης οδηγίας αναφέρεται αυτό. Επίσης ε, αναφέρεται ότι η νομοθεσία πρέπει να συνάδει με την ελεύθερη διακίνηση και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στη συνθήκη. Όλα λοιπόν πρέπει να συνάδουν με την προηγούμενη οδηγία. Η κυρία Χάνσλικ έχει επίσης κάποιες αμφιβολίες σχετικά με την ε, εφαρμογή των κανόνων στη χώρα υποδοχής αν ο εργαζόμενος ε, δεν δηλώνει αποσπασμένος υπάρχει το θέμα του ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο. Η νομοθεσία της χώρας ε, ε, υποδοχής ε, πρέπει να ισχύει. Επίσης έχουμε και αμφιβολίες για τη μετάφραση του εγγράφου. Το ιδεώδες για τη συνάδελφο θα ήταν να μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Όμως όταν είναι μακροσκελή τα κείμενα, η μετάφρασή τους μπορεί να δημιουργήσει εμπόδιο στην παροχή υπηρεσιών και αυτό δεν θα ήταν αποδεκτό. Τέλος, η συνάδελφος θεωρεί ότι είναι απόλυτα αναγκαίο να διευκολύνουμε την πρόσβαση στην ενημέρωση για την απασχόληση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση συλλογικών συμβάσεων, οι οποίες είναι δεσμευτικές και πρέπει να κοινοποιούνται και να είναι προσιτές, προσπελάσιμες και πρέπει να υπάρχει και συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και να προσδιοριστεί η σχέση μεταξύ χώρας αποστολής, χώρας υποδοχής. Για τα μέτρα ελέγχου λοιπόν, ο ρόλος αυτών των δύο χωρών είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου μόνο η χώρα υποδοχής ή η χώρα προέλευσης μπορεί να ε, έχουν σημασία. Χρειάζεται λοιπόν προσεκτική συνεργασία μεταξύ των δύο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και σας ευχαριστώ και εξ ονόματος ε, της συναδέλφου. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και την κυρία Χάνσλετ για την ξεκάθαρη θέση που εξέφρασε. Ε, ο κύριος ε, Πουζόη. Thank you very much, Chairman. Oh, uh, sorry. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη. Ε, τον κύριο Κοφεράτη ήθελα να πω. Εγώ φταίω. Κύριε Κοφεράτη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ε. Μπορεί να μιλήσει κάλλιστα πρώτος ο συνάδελφος. Σημασία έχει να μπορέσω να μιλήσω κι εγώ. Ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν την ε, συνάδελφο του Ρούνεν για όσα έχει κάνει, διότι πρόκειται για πολύ ευαίσθητη και δύσκολη δουλειά και έκανε τη δουλειά τη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εμεί ε, ω ομάδα συμμεριζόμαστε σε μεγάλο βαθμό την ε, τοποθέτησή της για το συγκεκριμένο θέμα και οι τροπολογίε που παρουσιάσαμε ω στόχο είχαν ε, και ελπίζω να τον επέτυχαν, να συνεισφέρουν στην ενίσχυση της γνωμοδότησης και να καθορίσουμε λίγο καλύτερα κάποιες συγκεκριμένε πτυχές. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για μας είναι σημαντικό κάποιες από τις λύσεις ε, που ανέφερε προηγουμένως η συνάδελφος να παραμείνουν και να γίνουν σεβαστές. Καταρχάς, ε, το να έχουμε ένα ανοιχτό κατάλογο στο άρθρο 3. Είναι σημαντικό να παραμείνει ανοιχτός αυτός ο κατάλογος, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να επιλέξουν και κάποια επιπλέον ε, κριτήρια ή κάποια κριτήρια τα οποία είναι μερικώς διαφορετικά από αυτά τα οποία έχουν καθοριστεί αρχικώς, ώστε να μην αποκλείεται κανένας, να μπορούμε να καλύψουμε όλες τις περιπτώσεις. Επίσης, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υιοθετηθούν κάποια κριτήρια. Ε, αναφέρθηκε, ε, για παράδειγμα, το τιμολόγιο και αριθμός των ε, συμβάσεων που συνάπτονται. Για μας αυτό είναι σημαντικό, ιδίως για την προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα παρόλα αυτά, με μια συγκεκριμένη οδηγία, χωρίς αυτό βέβαια ε, να δυσχεραίνει τη δυνατότητα να εφαρμόζονται συγκεκριμένα κριτήρια μέσω της ε, τιμολόγησης της εταιρείας και των συμβάσεων που συνάπτει κάθε επιχείρηση. Επίσης για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και για λόγους ε, σαφήνειας σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, να υπάρχει κάποια βεβαιότητα για τους ενδιαφερόμενους εργαζομένους και να μπορεί να καλύπτονται από την νομοθεσία ε, του κράτους μέλους που τους φιλοξενεί. Αν είναι καλύτερες οι προϋποθέσεις ε, στην ε, οικία νομοθεσία, τόσο το καλύτερο. Αλλά δεν θέλουμε να υπάρχει παρέκκληση από αυτό το στοιχείο βεβαιότητας. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να σας το πω, διότι θα πρέπει ευθύ εξ αρχή να διασφαλίζουμε ένα πλαίσιο αναφορά για του εργαζομένου, το οποίο να είναι κατάλληλο και επίση να είναι συγκεκριμένο και να μην αλλάζει συν το χρόνο. Ε, είναι πολύ καλέ οι προτάσει για την εφαρμογή των ελέγχων. Θα πρέπει από εκεί και πέρα την αρμοδιότητα για αυτούς τους ελέγχους να την έχει το κράτος ε, απόσπασης. Το άλλο κράτος θεωρείται ως ε, ε, θεωρείται υποκείμενο συνεργασίας, αλλά η ευθύνη θα πρέπει να είναι του κράτους απόσπασης. Επιπλέον, θα ήθελα να προσθέσω σε αυτές τις ε, σκέψεις και στα διάφορα σημεία τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και κατά την κατάθεση των συμβαστικών τροπολογιών, ότι αυτό το πιστοποιητικό δεν θα πρέπει να είναι το μόνο κριτήριο για να καθορίσουμε ότι μία επιχείρηση έχει έδρα σε μία χώρα ή όχι. Θα πρέπει να είναι ένα εκ των ε, ε, κριτηρίων, γιατί αυτό το ενιαίο πιστοποιητικό είναι προαιρετικό, δεν υποχρεώνει να υπάρχουν συγκεκριμένες ε, ενδείξει για μια επιχείρηση και αν υπάρχουν διαφορέ μπορεί να βρεθούμε ενώπιον τη εξή κατάσταση. Να έχουμε ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν καμία ευθύνη και να έχουν βρεθεί, να έχουν περάσει από τη μία χώρα στην άλλη και να ανήκουν σε διαφορετική εταιρεία, γιατί δεν προβλέφτηκε αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο στον καθορισμό της σχέση εργασία του. Τώρα, για τι διμερείς συμφωνίε που υπενθύμησε η συνάδελφο. Ε, είναι πολύ σημαντικό να περάσουμε στο σύστημα IMI. E Αλλά ακόμα δεν είναι σαφές πώς θα λειτουργήσει και πότε θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα IMI. E Επομένως, θα πρέπει να βρούμε μια λύση η οποία θα μπορέσει να μας εγγυηθεί, με τη δέουσα προσοχή βέβαια, και μια μετάβαση που δεν θα διακυβεύει τις διμερείς συμφωνίες. Θα ήθελα να προσθέσω επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν προσωρινά κέντρα ενημέρωσης ε, για τις διαβουλεύσεις αυτές, ώστε ένας αποσπασμένος που προέρχονται από δύο ή περισσότερους ανθρώπους που παρέχουν υπηρεσίες. Ε, υπάρχει ένας διτός ρόλος εδώ στο συγκεκριμένο θέμα και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη γιατί θα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ό,τι είναι σήμερα. Και επίση, Χρειαζόμαστε ένα σύστημα συνεχούς πληροφόρηση, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ώστε να μην εκθέτουμε σε περιτούς και αντιπαραγωγικού κινδύνους και τον ίδιο τον εργαζόμενο και την επιχείρηση, ιδίως σε περιπτώσεις στις οποίες ε, λόγω έλλειψης πληροφοριών και διαφάνειας μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. Στο τέλος άφησα γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, αλλά πρέπει να το λύσουμε και αυτό, το θέμα της ε, αλυσίδας υπεργολαβιών. Είναι ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει στην οδηγία για τις ε, δημόσιες συμβάσεις, αλλά ισχύει και για τις ιδιωτικές συμβάσεις. Θα έλεγα μάλιστα ότι σε αυτή την περίπτωση ε, θα έχει δεσπόδουσα θέση, κυρίως για τις ιδιωτικές συμβάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια λύση γνωρίζοντας ότι δυστυχώς στη μακριά αλυσίδα των συμβάσεων, βέβαια στην άλλη οδηγία θα προσπαθήσουμε να τη μειώσουμε αυτή την αλυσίδα, τουλάχιστον για τις δημόσιες συμβάσεις, αλλά δυστυχώς αυτή η αλυσίδα γίνεται όλο και μεγαλύτερη και όσο μεγαλύτερη γίνεται, τόσο μεγαλύτερη είναι η κίνδυση για τον ενδιαφερόμενο. Συνήθω οι καταχρήσει δεν γίνονται από τον πρώτο με τον οποίο συνάπτει κάποιο μια σύμβαση, αλλά με τον πιο απομακρυσμένο. Επομένω, θα πρέπει να αποφύγουμε αυτή η μακρά αλυσίδα να γίνει δομικό στοιχείο του μηχανισμού απόσπασης των εργαζομένων η συνάδελφος αναφέρθηκε σε αυτό. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα, το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε με τη δέουσα προσοχή, αλλά πρέπει να βρεθεί μια λύση και για αυτή την πτυχή. Κατά τα λοιπά, ε, πρέπει να δούμε τι ακριβώ μα λείπει προκειμένου να καταλήξουμε σε καλέ συμβαστικέ προτάσει. Αλλά εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο για τη δουλειά τη. Ε, έδειξε ιδιαίτερο πάθος, αλλά κατάφερε ταυτόχρονα να λύσει και μέχρι τώρα με πολύ επαγγελματικό τρόπο σημαντικά ζητήματα. Thank you very much indeed, Mr. Kofarati. Uh, now, Mr. Bezoy. Thank you, President. Uh, I would like to be brief and uh, make a few remarks on those aspects of the proposed directive which are of great importance. I refer to Articles 3, 6, 9, 12,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 δεν πρέπει να καταλήξουμε ε, σε διαφορετικά συμπεράσματα ανάλογα με το κράτος μέλος και ε, τις καταστάσεις. Δεν θα πρέπει να είναι η προσέγγιση μας, πιστεύω. Σχετικά τώρα με την πρόταση της Επιτροπής για το άρθρο 9, μέτρα ελέγχου, ε, αυτό θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε νέα κριτήρια, αν παραστεί ανάγκη. Για τα κριτήρια τώρα, είμαι υπέρ της διαγραφής του τελευταίου σημείου, το οποίο αναφέρεται σε περιορισμένο αριθμό fashion στο κράτος μέλος εγκατάστασης. Στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων, κυρίως στην περίπτωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εάν υπάρχει μια σύμβαση στο εξωτερικό, είναι διαφορετικό. Για μια δεδομένη χρονική περίοδο είναι φυσιολογικό να συμβεί αυτό σε ένα κράτος μέλος και όχι στο κράτος μέλος εγκατάστασης. Γι' αυτό το λόγο δεν πρόκειται πάντοτε για αυτή μια τέτοια περίπτωση. Όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τους όρους, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να διευκολύνουμε την πρόσβαση στις πληροφορίες σε, ε, σε εκείνους ε, που παρέχουν τις υπηρεσίες κυρίως όταν πρόκειται για συλλογικές συμβάσεις, αν θέλουμε να διευκολυνθεί η απόσπαση των παρόχων υπηρεσιών. Οι παρόχοι υπηρεσιών πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για να γνωρίζουν από την αρχή τι πρέπει να κάνουν ε, με τους υπαλλήλους τους. Δεν γνωρίζω αν η δημιουργία κέντρων, προσωπικών κέντρων ενημέρωση θα λειτουργήσει όπως προτείνεται τις ορισμένε τροπολογίες. Δεν ξέρω αν αυτό δεν θα είναι ένα επιπλέον βάρος και όχι μια προστιθέμενη αξία για τους αποσπασθέντες για τη Γενική Αρχή της Αλληλοβοήθειας αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συμφωνώ υπέρ της αμοιβαίας βοήθειας, αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια ρεαλιστική προθεσμία για τα κράτη-μέλη. Δηλαδή ένας εύλογος χρόνος για να μπορεί να αντιδράσει κανείς σε ένα άλλο κράτος μέλος. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε εδώ την πρακτική. Νομίζω ότι η προθεσμία που προβλέπει η Κομισιόν είναι στενή. Γι' αυτό το λόγο προτείνω μια προθεσμία 30 ημερών. Αυτό θα συζητηθεί βεβαίως. Ε, άλλοι συνάδελφοι αναφέρονται για ένα μήνα ε, για τους μηχανισμούς ε, ε, επίγοντες μηχανισμούς. Για ορισμένα κράτη-μέλη αυτή η πρόταση δεν είναι ρεαλιστική. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μία, δύο ή τρεις εργάσιμες ημέρες. Δεν θα αλλάξουν πολλά για την ε, δηλούς αρχή, αλλά τουλάχιστον το άλλο κράτος μέλος θα έχει χρόνο να αντιδράσει. Άρθρο 9. Μέτρα ελέγχου. Επιμένω επί της ανάγκης να υπάρχει μια ε, λεπτομερής λίστα για να υπάρχει ενιαία προσέγγιση. Στην Ένωση με άλλους συναδέλφους προτείναμε αντίγραφο της ε, Σύμβασης Εργασίας Απασχόλησης είτε ηλεκτρονικό αντίγραφο είτε ε, σε χαρτί για το άρθρο 12. Uh, το τελευταίο σχόλιο που θέλω να κάνω σχετικά με την ευθύνη, αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, αντιλαμβάνομαι ότι ορισμένα συστήματα λειτουργούν πολύ καλά σε κράτη-μέλη, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε μια λύση σε κοινωτικό επίπεδο. Τώρα, εάν κάποιος τηρεί αυτή την υποχρέωση, πρέπει να αναλαμβάνει και την ευθύνη. Αυτό είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει το δικαστικό σύστημα. Και δεν βλέπω για ποιο λόγο ο συμμελόμενος είναι ε, ο αναθέτων είναι υπεύθυνο όταν η συμβαλώνει και οι συμβαλώνει και οι υπεργολάβοι δεν τηρούν τις ευθύνες τους. Χρειάζεται να υπάρχει αμοιβαία ευθύνη. Αν όμως δεν υπάρχει ορισμός, καθορισμός της δέουσας επιμέλειας, νομίζω ότι αυτό δεν θα λειτουργήσει. Προτείνω τα κράτη-μέλη που θέλουν να δημιουργήσουν ένα τέτοιο σύστημα, που θα είναι σύμφωνο με το δικαστικό σύστημα, προτείνω να μπορούν να το κάνουν. Δεν νομίζω να πρέπει να επιβάλλουμε αυτό το σύστημα σε όλα τα κράτη-μέλη και κυρίως όχι ε, σε, όλους, ε, σε όλη τη γραμμή υπεργολαβίας. Γι' αυτό το λόγο, κατά τη δική μου άποψη, το μόνο το οποίο μπορεί να συμβεί είναι να αποθαρρύνουμε ε, τις επιχειρήσεις ε, που θα φοβηθούν ότι με τους αποσπασθέντες θα έχουν μεγαλύτερο βάρος. Βεβαίω είμαι έτοιμο να συζητήσουμε και πάντοτε με διάθεση να βρεθεί ένα συμβασμό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μιλήσω εκ μέρου τη ομάδα μας ως... Ε, Build, uh, on what a number of colleagues... Ε, υπόψη και αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, νομίζω ότι από τη δική μα την προοπτική Καταλαβαίνουμε και δεχόμαστε ότι πρέπει να βελτιώσουμε την επιβολή στην οδηγία για την απόσπαση. Ε, αργότερα θα συζητήσουμε και για την οδηγία των υπηρεσιών και την εφαρμογή της και αυτό είναι ενδιαφέρον σε αυτό το πλαίσιο. Όταν ψηφίσουμε για την οδηγία για τις υπηρεσίες θα το συνδέσουμε με μία ενθάρρυνση ε, στην Κομισιόν να προωθήσει και την οδηγία για την απόσπαση. Αυτές οι δύο οδηγίες κινούνται παράλληλα, γιατί η οδηγία για την απόσπαση αναμφίβολα συνδέεται με το όλο θέμα της ελευθερίας εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών. Και θα πρέπει η ενιαγορά να δουλέψει καλύτερα μέσα από την καλύτερη επιβολή των μέτρων της νομοθεσίας. Η εστίαση λοιπόν της νομοδότησης της Επιτροπής μας αυτή πρέπει να είναι. Δεν είναι ευκαιρία αυτή για να τροποποιήσουμε ή να αλλάξουμε το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Έτσι λοιπόν εξετάσαμε και συνυπογράψαμε αρκετές προτάσεις των συναδέλφων για να διασφαλίσουμε ότι η οδήποτε μέτρο ε, υιοθετηθεί δεν θα δημιουργεί διακρίσεις δεν θα δημιουργεί άχρηστο διοικητικό φόρτο και δεν θα αποθαρρύνει ενεργά τον κόσμο από το να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δίνει η οδηγία ε, για τι ενιαία αγορά για τι υπηρεσίε. Και ιδιαίτερα δεν πρέπει να αποθαρρύνουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα στην αγορά εργασία. Θέλουμε να δημιουργηθούν θέσει εργασία, να ανοίξουν νέε ευκαιρίε αυτός ήταν ο σκοπός της ε, αρχικής οδηγίας για τις υπηρεσίες που την τροποποίησαμε ώστε όλα αυτά να είναι σωστά. Κάναμε λοιπόν προτάσεις για το άρθρο 3, υπ' αυτή την έννοια που σας περιέγραψα, που είναι πολύ ρεαλιστικές προτάσεις πιστεύουμε. Επίσης το 7, 5 και 9 για να υπάρχει καλή ισορροπία μεταξύ της σωστής επιβολής αλλά χωρίς ε, αποτρεπτικό φόρτο και διοικητικό φόρτο στις μικρές ΜΜΕ. Επίσης το σύστημα πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς, ε, το IMI, ε, είναι πολύ σημαντικό για την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες και οι αρμόδιες αρχές έτσι θα μπορούν να συνεργάζονται να ε, δίνουν την έγκρισή τους όπου αυτή χρειάζεται σε τοπικό επίπεδο. Οι αρμόδιες αρχές πραγματικά έχουν κέριο ρόλο εδώ να παίξουν. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αν δεν δώσουμε κάποια κίνητρα το σύστημα IMI δεν θα χρησιμοποιείται. Ενώ ο σκοπό του είναι να χρησιμοποιείται για να βελτιώνονται όλες αυτέ οι διασυνοριακές ε, συναλλαγές. Τέλο, συμφωνούμε, και το είπε και ο κύριος ε, Μπουζόη, δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιβάλλουμε συγκεκριμένη διατύπωση όπως ε, συστήματα ευθύνης ε, εξ και από κοινού, κοινού και εις ολόκληρων. Επίσης, ε, το ίδιο θέμα θα προκύψει και στις δημόσιες συμφάσεις το θέμα της επιβολής και η ποιότητα της επιβολής της οδηγίας απόσπασης είναι διαφορετικό και το πώς αντιμετωπίζεται η αγορά εργασίας είναι διαφορετικό. Εδώ υπάρχουν κάποια εργαλεία που ίσως δεν εξυπηρετούν όλους. Είμαστε ανοιχτοί να συνεχίσουμε τη συζήτηση με την Έμιλη Τούρουνεν και πιστεύω ότι θα επιτύχουμε κάποιες καλές συμβαστικές λύσεις που θα επικεντρώνονται στο θέμα ε, της ε, δικής μας επιτροπής, ε, γιατί εμείς ε, έχουμε ασχοληθεί πολύ με την οδηγία για τις υπηρεσίες και ξέρουμε και τα παράλληλα θέματα μεταξύ των δύο οδηγιών. Μπορούμε λοιπόν να συζητήσουμε και με την Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή και η Επιτροπή Απασχόλησης θα υποβάλει, ε, πιστεύουμε, καλές προτάσεις. Και ο κύριος Χάντλ τώρα. Να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή αναλάβατε από τον κύριο Γκούσταυσον ως ε, τακτικό μέλος της Επιτροπής μας. Με χαρά σας καλωσορίζουμε και με χαρά σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για το καλωσόρισμα. Ε, συγγνώμη που την περασμένη φορά την προηγούμενη φορά όταν μιλάγαμε για το προηγούμενο θέμα δεν πήρα το, το λόγο. Δεν ε, είμαι εξοικειωμένος με τις ε, συνήθειες κάθε επιτροπής, σε μια άλλη επιτροπή είναι διαφορετικές ε, οι συνήθειες. Η συνάδελφος του Ρούνεν υπέβαλε εξαιρετική έκθεση και έκανε και εξαιρετική προετοιμασία για τις περαιτέρω εργασίες μας. Ε, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό γιατί τη γνωρίζω από τη συνεργασία μας στην Επιτροπή Απασχόλησης. Ευχαριστώ θερμά λοιπόν Έμιλη. Νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι ένα αντικείμενο που επιβεβαιώνει ότι όσο περισσότερο προσπαθούμε να επέμβουμε ρυθμιστικά νομοθετικά σε, για να λύσουμε διάφορα προβλήματα ή θέματα, τόσο ταχύτερα αναπτύσσεται το θέμα της καταστρατήγησης των διατάξεων που θέτουμε το θέμα της ε, παροχής υπηρεσιών και της απόσπασης είναι σημαντικές διατάξεις που δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ και 20 χρόνια έχω πείρα πρακτικής δουλειάς ως γραμματέας ε, ε, του συνδικάτου στις επιχειρήσεις και τώρα ακόμα έχω επαφή με πολλούς εκπροσώπους συνδικαλιστικών συμφερόντων αλλά και εργοδοτικών συμφερόντων που όλοι μου παραπονούνται για την καταστρατήγηση των διατάξεων που έχουμε ε, θεσπίσει για τη ρύθμιση. Δεν πρόκειται μόνο για τις προϋποθέσεις των αποσπασμένων ε, εργαζομένων, αλλά και τις προϋποθέσεις των εργοδοτών στον τόπο εγκατάσταση, στην επιχείρηση, μισθολογικό ντάμπινγκ. Βεβαίως πρόκειται και για το θέμα του δίκαιου και θεμητού ανταγωνισμού και των συνθήκων ανταγωνισμού και σε σχέση με το τοπικό εργατικό δυναμικό, το οποίο πολλές φορές παραπονείται πικρά για το dumping ε, από επιχειρήσεις ε, άλλων κρατών μελών που προσπαθούν να βρουν καλύτερες ε, ε, προϋποθέσεις ε, και με μισθολογικό dumping να καταστρατηγήσουν την υφιστάμενη νομοθεσία. Άρα λοιπόν πρέπει να ρυθμιστεί σωστά το θέμα. Εγώ θα επισέλθω σύντομα σε τρία ζητήματα. Νομίζω ότι κάθε ρύθμιση νομοθετική από την πλευρά μας ε, θα στερείται νοήματος και αξίας αν δεν έχει επαρκή έλεγχο, δυνατότητα ελέγχου και αν δεν έχει επαρκείς κυρώσεις. Ε, πολλές φορές ε, μιλάμε για υπερβολική γραφειοκρατία, αλλά εδώ θέλει προσοχή, μην κάνουμε λάθος, γιατί οποιαδήποτε νομοθεσία ε, που δεν υπόκειται σε έλεγχο και σε κυρώσεις, σε τελευταία ανάλυση δεν αξίζει τίποτε, διότι ε, γίνονται συχνά καταχρήσεις και καταστρατηγήσεις ατιμωρητοί. Δεύτερον, Νομίζω ότι είναι σημαντικό σε σχέση με το θέμα της ε, ευθύνης, ε, δηλαδή ε, από κοινού και ισολόκληρων, εκεί πρέπει να βρούμε μια διατύπωση, ούτω ώστε να ρυθμίσουμε τα θέματα αυτά της καταστρατήγησης, γιατί από την έκθεση πολλών εργοδοτών, από εκθέσεις πολλών εργοδοτών, γνωρίζω ότι οι εργαζόμενοι πολλές φορές γνωρίζουν ότι ε, ο επόμενος υπεργολάβος δεν θα τηρήσει τις ε, προϋποθέσεις για την εργασία, συλλογικές συμβάσεις κλπ. Και αυτό πρέπει να το εμποδίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν λέω ότι αυτό είναι ο κανόνας, αλλά σε πολλές περιπτώσεις γίνονται συστηματικές ε, καταχρήσεις για να... και καταστρατηγήσεις. Τέλος, η, η συγγήτρια αναφέρθηκε και στην κυρία Χάνσλιγκ. ελπίζω αυτό που θα πω να το κατάλαβα λάθος, διότι εμείς ε, δεν μπορούμε ε, να στηριζόμαστε στις απαγορευτικές αποφάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αν το δικαστήριο λαμβάνει μια απόφαση με βάση τις μέχρι τούδε ε, οδηγίες ε, και νομοθετήματα και θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τότε είναι καθήκον μας να προβούμε σε τροποποιήσεις, ούτω ώστε οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι να μπορούν να λειτουργούν με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις σε κάθε χώρα. Αυτό έχει να κάνει με τη διαφάνεια, έχει να κάνει και με τον έλεγχο και προς εκεί πιστεύω ότι πρέπει να κινηθούμε και να συμφωνήσουμε στην έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, και οι επόμενες παρεμβάσεις σας θα είναι ευπρόσδεκτες. Άλλα μέλη, μη σκιώδης, ο κύριος Ομπερμάγερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταλαβαίνω αυτό που είπατε ότι πρέπει αφενός να κρατήσουμε χαμηλά το γραφειοκρατικό φόρτο αλλά από την άλλη και το υπογραμμίζω αυτό να υπάρχει ασφάλεια δικαίου, προστασία εργαζομένων, θεμητός ανταγωνισμός για τις ε, ντόπιε επιχειρήσεις στη χώρα υποδοχής. Όλα αυτά πρέπει όπως πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και να βρούμε την ισορροπία μεταξύ των δύο ομάδων συμφερόντων. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα από αυτά που συζητήθηκαν που έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα ελέγχου των αρχών είτε στη Γερμανία είτε αρχές σε άλλες χώρες. Ε, να αναφέρω κάποια θέματα που χρήζουν συζήτηση. Ένα σημαντικό θέμα που αναφέρθηκε ήδη είναι η δυνατότητα ελέγχου των εγγράφων. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτονόητο να γίνει ένας σοβαρός έλεγχος της, ε, ε, των, των ε, δελτίων μισθοδοσίας και άλλων στοιχείων που δείχνουν τον, το είδος της απασχόλησης. Αυτά θα πρέπει να τεκμηριώνονται και να υπάρχει δυνατότητα εξέτασης όλων των σχετικών εγγράφων. Η επίδοξη διαβατηρίου ή κάποιου άλλου παρομοίου γράφου ταυτότητας. Και αυτό είναι σημαντικό. Έχει να κάνει με τη διαφάνεια. Ε, επίσης είναι ε, ε, σημαντικό να δούμε και τον ρόλο του εκπροσώπου των εργαζομένων που δεν προβλέπεται γιατί είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος αυτός για να αντιμετωπίσουμε διάφορα περίπλοκα προβλήματα. Ε, επίσης, ε, γιατί δεν θα πρέπει να γίνεται μια αμερόληπτη εξέταση για να εξετάσει και τους κινδύνους που ε, εξαρτώνται από την επιχείρηση και την εργασία, ε, όπως και είναι, είναι σημαντικό επίσης να λαμβάνεται υπόψη και ο αριθμός των εργαζομένων. Ανεξάρτητα όμως από το αν πρόκειται για 5 ή 10 ή 500 θυγόμενους εργαζομένους, πιστεύω ότι θα πρέπει παρόλα αυτά να γίνεται έλεγχος. Επίσης, ό,τι δεν ε, αντιμετωπίζεται με κυρώσεις ε, δεν έχει καμία αξία. Θα πρέπει λοιπόν οι κυρώσεις να μπορούν να εκτελούνται και να εξασφαλίζουμε τη δυνατότητα εκτέλεσης των ε, κυρώσεων που προβλέπονται σε κάθε κράτος μέλος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Κομισιόν παρακολουθεί, δεν ζήτησε το λόγο. Υπάρχει και μια ομάδα εργασίας του Συμβουλίου ε, σήμερα. Η κυρία Φίνστρο που είναι υπεύθυνη δεν είναι εδώ. Ε, δεν ζητεί το λόγο. Δεν ζητεί. Ακούει όμως. Κυρία Τούρινεν, να σας δώσω το λόγο για να συνοψίσετε την κατάσταση των πραγμάτων, να μας πείτε για τα χρονοδιαγράμματα και ό,τι άλλο θέλετε. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν στη συζήτηση. Είναι κάτι το ενδιαφέρον και νομίζω ότι φτάνουμε σε ουσιαστικά προβλήματα και θέματα. Τώρα για το ΕΛΚ. Νομίζω Παρακαλώ να πείτε στην κυρία Χανσλίκ ότι δεν βρισκόμαστε απαραίτητο τόσο μακριά ημένα από τους δε. Ίσως ε, το ξεκίνημα, η αφετηρία μας είναι διαφορετική, ναι. Αλλά νομίζω, ως προς τα περισσότερα άρθρα, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε. Για το άρθρο 9. Εξ ονόματος κυρία Χάνσλιφ, είπατε ότι σημαντικό είναι για εσά να βελτιωθεί η νομική ασφάλεια και να υπάρχει ένα κλειστός κατάλογος. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακούσουμε και τις εθνικές αρχές, τους ειδικού, επειδή ζητούν λίγο περισσότερη ευελιξία. Από την άλλη πλευρά, όπως είπα, μπορούμε να δημιουργήσουμε και μεγαλύτερη διαφάνεια σε κάθε κράτος μέλος πως είναι εύκολο να δούμε ποιο θα είναι το ζητούμενο από την κάθε επιχείρηση, τι περιμένουμε από την κάθε επιχείρηση. Επίσης, ε, η κάθε, να υπάρχει υποχρέωση να δημοσιεύονται τα εθνικά μέτρα ελέγχου. Υπάρχουν, θα υπάρχουν φυσικά μικροδιαφορές μεταξύ των κρατών μελών και θα μπορούσε να υπάρξει ένας πυρήνας ευρωπαϊκός, μια βάση ευρωπαϊκή, ε, που θα είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη-μέλη. Ας προσπαθήσουμε να τα δούμε περισσότερο. Επίσης, βλέπουμε ότι ο οικονομικός κλάδος απασχολεί πολλούς και μάλιστα είμαστε, είναι, η οργάνωση των εργοδοτών είναι υπέρ μιας ανοιχτής λίστας. Θα πρέπει να δούμε την πρακτική πλευρά του θέματος και να το εξετάσουμε περισσότερο. Επίσης, το ΕΛΚ ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, πιο εύκολη πρόσβαση στην πληροφόρηση, συμφωνώ απόλυτα. Εδώ μπορούμε να προχωρήσουμε, πιστεύω και σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και για τις επιπλέον τροπολογίες σας. Ορισμένες παρατηρήσεις είναι σωστές και πρέπει να περιληφθούν ε, στις συμβαστικές προτάσεις. Για το Άλντε, για το άρθρο 3, πάλι ο κ. Σόγια μίλησε για την νομική ασφάλεια και για ε, την σαφήνεια των ορισμών πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες από το κλείσιμο μιας λίστας. Μπορεί να υπάρχει δυνατότητα να παρεκκλίνει κανείς από αυτήν. Ίσως πάλι μια λύση θα ήταν να υπάρχει ένας πυρήνας, αλλά ας το εξετάσουμε περισσότερο. Πάλι για το θέμα της πληροφόρησης, της ενημέρωσης, συμφωνώ για το χρόνο, ναι, είναι πρακτικό. Για την κοινή ευθύνη. Πολλοί το ανέφεραν. Αυτό το θέμα είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι υπάρχει μια, ένας κατακαιρματισμός στην ενιαία αγορά, διότι οκτώ μέλη έχουν δημιουργήσει μια κοινή υπευθυνότητα και συνεπώς ορισμένα ε, μία χώρα θα έχει ένα σύστημα, όπως τη Γερμανία, μια άλλη χώρα θα έχει άλλο σύστημα και μια τρίτη χώρα ένα τρίτο θέμα. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω ότι δυστυχώς υπάρχει κατακαιρματισμός σήμερα και θα έπρεπε να έχουμε ένα κοινό ορισμό εισόφλησης ενιαίας αγοράς και κατόπιν να δούμε αυτή την ε, επιμέλεια ε, διότι εάν έχετε κάνει όλους τους ελέγχους, τελικά δεν μπορείτε να ζητήσετε κατά πόσο είναι πλαστά τα έγγραφα. Υπάρχει, υπάρχουν όρια στα, στο τι περιμένετε. Τελικά μπορεί να το ψηφίσουμε αυτό, αλλά ας δούμε τι θέλουν τα διάφορα κράτη-μέλη. Ένα άλλο θέμα αναφέρεται ότι οι αγορέ εργασία στην Ευρώπη διαφέρουν, συμφωνούμε. Συνεπώ πρέπει να βρεθεί ισορροπία, να υπάρχει ορισμένη ευελιξία στο εθνικό επίπεδο, αλλά η ευρωπαϊκή αγορά εργασία ενοποιείται κατά κάποιον τρόπο. Όλο και περισσότερα άτομα είναι αποσπασμένα και γι' αυτό χρειάζεται ένα κοινό έδαφος και για να δημιουργηθεί αυτό το κοινό έδαφος πρέπει να συνεισφέρουμε ενεργά. Νομίζω ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχει διαφορά, τουλάχιστον στη χώρα μου και σε άλλες χώρες, υπάρχει διαφορά μεταξύ μεγάλων ε, επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων. Μεγάλη διαφορά. Επειδή οι μικρότερες επιχειρήσεις είναι εκείνες ε, οι οποίες χάνουν από πλευράς ανταγωνισμού όταν δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Όταν υπάρχουν ορισμένε επιχειρήσεις που δεν τηρούν τους εθνικούς κανονισμούς ε, Στη Δανία, για παράδειγμα, βλέπω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που χάνουν και οι μεγάλες είναι εκείνες που κερδίζουν όλα τα χρήματα διότι έχουν έναν ξένο υπεργολάβο που στέλνει αποσπασμένου εργαζόμενου και τελικά οι μεγάλε επιχειρήσει είναι εκείνε που κερδίζουν τα περισσότερα. Και αυτό αφορά και τι ε, ξένε επιχειρήσει και του ε, αποσπασμένου. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει και πρέπει να υπάρχει ένα σωστό υγιή ανταγωνισμό μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων. Για την ΚΟΥ ευχαριστώ πολύ. Συμφωνούμε σε πολλά σημεία και είναι αυτό που είπατε, το πρακτικό θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία σας από την γερμανική αγορά εργασίας. Τέλος, για τη διαδικασία. Σήμερα θα υπάρξει μια συνεδρίαση του προσωπικού και κατόπιν έχουμε δύο συνεδριάσεις τις ερχόμενες εβδομάδες ε, των σκιωδών συντονιστών. Θα έχουμε δύο. Ε, η δυσκολία είναι να βρούμε αίθουσες και διερμηνία, αλλά νομίζω θα τα καταφέρουμε και θα εστιάσουμε στα βασικά θέματα και ελπίζω ότι θα υπάρξουν ήδη πολλά άρθρα από την οποία θα συμφωνήσουμε στις δύο πρώτες συνεδριάσεις των σχεδόν συντονιστών και κατόπιν θα ψηφίσουμε εδώ σε αυτή την Επιτροπή. Ίσως θυμάστε καλύτερα, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Νομίζω το Δεκέμβριο και μετά στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου. Δεν θυμάμαι πολύ καλά τις ημερομηνίες. Ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ πολύ. και νομίζω ότι η ικανότητά σας θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε καλά αποτελέσματα. Τώρα πρόκειται να το υιοθετήσουμε στις 18 Δεκεμβρίου και κατόπιν στις 18 Φεβρουαρίου τον Ιανουάριο θα γίνει μια μεγάλη ψηφοφορία που γνωρίζουμε 18 Δεκεμβρίου θα γίνει η ψηφοφορία και ελπίζω ότι μέχρι τότε θα έχετε μια συμβαστική πρόταση. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα σε μια άλλη σημαντική γνωμοδότηση. Είναι ε, μια νέα πρόταση για την προστασία των φυσικών προσώπων ενάντια της επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό για να λειτουργήσει η νέα αγορά. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον υπήρξε για αυτή τη γνωμοδότηση. Έχουμε 159 τροπολογίες ε, που δείχνουν το ενδιαφέρον των μελών και σας ευχαριστώ όλους γι' αυτό. Η συγγήτριά μας είναι η κυρία Κόμη, η οποία είναι παρούσα. Επίσης, η κυρία Σαντεμούσα, ο κ. Άγκστρον, νομίζω, εγώ είμαι συνσηγητής ε, με την κυρία Λίμπερς, η κυρία Γκάλο είναι παρούσα. Είσαστε επικεφαλής συσυχήτρια, νομίζω για αυτό το θέμα. Και... δεν είναι παρούσα, ο κ. Σαρδίν είναι εδώ. και οποιοδήποτε άλλο θέλει να μιλήσει. Έχουμε τον κύριο Γκάλο, κύριο Σαμπίτ, οποιοδήποτε θέλει να εγγραφεί στον κατάλογο μιλητών, ευχαρίστω. Μέχρι τι 12.30 μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα, δεν υπάρχει πολύ χρόνο. Αλλά παρόλα και γι' αυτό σα παρακαλώ να είσαστε όσο το δυνατόν πιο συνοπτικοί. Κατόπιν έχουμε και την Επιτροπή. Η κυρία Μπουλούντσε ναι, θα μιλήσει ε, εξ ονόματος της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης. Εντάξει. Παρακαλώ την κυρία Κόμη να μας παρουσιάσει ε, τις απόψεις της για τις ε, τροπολογίες της 156. Εσείς έχετε καταθέσει 7 νομίζω. Υπάρχουν πάνω από 300 τροπολογίες. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να βρούμε το δρόμο μας ώστε να υπάρχει τελικά μία γνωμοδότηση ισχυρή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως όπως είπατε το θέμα είναι πολύ περίπλοκο και Υπάρχει μια πολιτική δυναμική, αλλά ε, μας ενδιαφέρει και κοινή λογική. Γι' αυτό είναι και ο λόγος ε, που καταθέσαμε τόσες πολλές τροπολογίες. Θα προσπαθήσω να σας καθυστερήσω όσο το δυνατόν λιγότερο, αλλά πρέπει να διευκρινίσω οπωσδήποτε κάποια θέματα εδώ μαζί σας και μετά θα διευκρινιστούν και κάποια άλλα θέματα στη συνεδράση με τους κοιόδης συμπληκτές που θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που είναι εδώ, ε, διότι παρά το γεγονός ότι έχουμε απλώς μια γνωμοδότηση στην Επιτροπή μας, ε, είναι θεμελιώδους σημασία, διότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε το όλο σύστημα και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία διαπιστώσαμε ήδη. Θεωρώ ότι υπάρχουν οι βάσεις για να γίνει εξαιρετική δουλειά και να παραδώσουμε στη συνέχεια στην καθήλυνα αρμόδια επιτροπή μια ισορροπημένη και ακριβή γνωμοδότηση που θα αφορά τα πιο σημαντικά σημεία χωρίς να περιπλέκουμε τα πράγματα. Αυτό είναι ο κίνδυνος που ελοχεύει. Να μην επικεντρωθούμε αντικειμενικά στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς, αλλά ορισμένες φορές να επισέλθουμε και σε άλλα ε, μονοπάτια. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω και από τους συναδέλφους να ε, σταθούμε στα στενά όρια της Επιτροπής μας. Ζήτησα από την προηγούμενη εβδομάδα συνάντηση με τους κοιόδης εισηγητές για να προσπαθήσουμε να περάσουμε στην ουσία των διαφόρων θεμάτων παρά το γεγονό ότι η αρχική μου πρόθεση ήταν να επικεντρωθώ στα θέματα τα οποία είναι δική μα αρμοδιότητα, όπω είπα προηγουμένω, σέβομαι και το γεγονό ότι κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να τροποποιήσουν όλα τα κεφάλαια, ιδίω το κεφάλαιο που αφορά τη μεταφορά δεδομένων. Θα πρέπει καταρχάς να ξεκινήσουμε από τους ορισμούς. Θεωρώ ότι αυτό είναι το σημείο εκκίνωσης στην ε, παρούσα οδηγία είχαμε κάποιους ορισμούς που ήταν χρήσιμοι και μπόρεσαν να αντέξουν τις τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων 7 ετών, αλλά θα πρέπει ίσως να έχουμε και κάποιους ορισμούς και, ε, και ορολογία που θα είναι ε, κατάλληλοι για τα μέσα που χρησιμοποιούμε το 2012. Η βασικότερη πρόκληση θα είναι να αποφασίσουμε ποιες νομικές βάσεις μας επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα κάποιων και τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να δώσουμε τελικά στη συνένεση. Αυτό το οποίο θα πρέπει να λάβουμε λάβουμε υπόψη είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι απαιτήσει και η συγκεκριμένη μορφή μπορεί να αποτελέσουν ε, άχθος όσο και αν αυτό αφορά την ε, μεγαλύτερη δυνατή προστασία για τους καταναλωτές. Επομένως, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αυτόν τον κανονισμό, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι κυρίω μα ενδιαφέρει η προστασία του καταναλωτή. Θα πρέπει να έχουμε κάτι για να διασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ευολεξία, χωρί αυτό να είναι ει βάρο τη προστασία των ατόμων. Και αυτό είναι επίση σημαντικό. Και επίση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στι γενικέ αρχέ και την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν παιδιά ή και πιο ευάλωτε ομάδε που αναφέρονται στο άρθρο 9 και στο άρθρο 11 θα πρέπει να υπάρχει εκεί μεγαλύτερη προσοχή. Στα δικαιώματα τώρα. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με διάφορα στοιχεία. Καταρχάς, ε, οι τροπολογίες που κατατέθησαν ε, αφορούν κάποια γενικά μεν θέματα, αλλά υπάρχουν και κάποιες λεπτομέρειες. Παραδείγματος χάρη το δικαίωμα στην ενημέρωση, το δικαίωμα της ένστασης, αλλά τα πιο διαφιλονικούμενα ζητήματα είναι σίγουρα το δικαίωμα της διαγραφής, ε, της λήθης. Και επίσης το πώς επεξεργάζεται κάποιος τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Θα ήθελα να σταθώ λοιπόν σε αυτά τα στοιχεία. Το πρώτο από τα οποία ανέφερα είναι λογικό, αλλά αφορά κυρίως τον ψηφιακό κόσμο, στον οποίο ούτως ή άλλως θα πρέπει να κάνουμε προσαρμογές. Το δεύτερο που ανέφερα θα πρέπει να τη χάνει συγκεκριμένου νομοθετικού μέσου, ξεχωριστό, αφορά δηλαδή τη μεταφορά δεδομένων, δεδομένου ότι είναι πολύ περίπλοκο να το εφαρμόσουμε και είναι πολύ λίγη χρησιμότητά του στο συγκεκριμένο κανονισμό. Πρόκειται για ένα μέσο το οποίο ε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα όσον αφορά τα δικαιώματα του ατόμου και θα πρέπει να κατανοήσουμε αν η Επιτροπή μα, η ΙΜΚΟ, που κυρίω ενδιαφέρεται για την προστασία των καταναλωτών, προτιμά να υπάρχει καλύτερη διάρθρωση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπής ή θα έπρεπε να μείνει στα χέρια των ε, δικαιωμάτων των ε, ατόμων. Θα πρέπει να δούμε και προ ποια κατεύθυνση θέλουμε να κινηθούμε. Όσον αφορά την τελευταία ψυχή, ε, πτυχή, συγγνώμη, την κατάρτιση του προφίλ, θα πρέπει να δούμε τι νομικέ πτυχέ και τα πιο ουσιαστικά στοιχεία, διότι για το σημείο αυτό Κατά πάσα πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί ε, μία ορολογία η οποία δεν διευκρινίζει επακριβώς τις προθέσεις της και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε μια πολιτική κατεύθυνση που ε, θα διασκεδάσει αυτή τη νομική ασάφεια που διαπιστώσαμε στο κείμενο. Ο τέταρτος τομέας εργασίας αφορά τον έλεγχο και την επεξεργασία των δεδομένων. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάλογα με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του καθενός ε, ενώπιον και των ατόμων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν θα πρέπει η κάθε κατηγορία όμως να ε, τεθεί εντός ε, πολύ αυστηρών πλαισίων διότι διάφορες κατηγορίες περιλαμβάνουν αρκετά στοιχεία και θα, αυτό θα σημαίνει ότι θα μειωθεί ευελιξία. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση και το γνωρίζει αυτό η Επιτροπή μας. Θα πρέπει να μιλήσουμε και για το cloud computing, ε, να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι ε, το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα χάνει κάποιες ιδιότητες και γίνεται στην πραγματικότητα ο ελεγκτής και πρέπει να δούμε και τι γίνεται με αυτόν που επεξεργάζεται τα δεδομένα. Θα πρέπει να δούμε και τι όρια υπάρχουν μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου και μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να φτάσουμε για την προστασία των δεδομένων. Από εκεί λοιπόν ε, μας ενδιαφέρει κυρίως ο ορισμός του ατόμου στον οποίο φέρονται τα δεδομένα, αλλά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνουν τα πάντα εις βάρος της προστασίας, γιατί ο στόχος μας, επαναλαμβάνω, είναι να προστατεύσουμε τον καταναλωτό τον καταναλωτή. Επίσης μας ενδιαφέρει και το θέμα της κοινοποίησης της παράνομης ε, ή νόμιμης πρόσβασης στα δεδομένα και αυτό είναι σημείο κλειδί. Αρκετές πολιτικές ομάδες ε, θίγουν και το θέμα της εφαρμογής ε, αυτής της προθεσμίας των 24 ωρών, αλλά οι διάφορες εναλλακτικές λύσεις που προτείνονται δεν μας επιτρέπουν προς το παρόν να κατανοήσουμε αν θα υπάρχει ρητή μνήα στο συγκεκριμένο όρο ή θα ε, επικεντρωθούμε στην κοινή μας λογική. Όσον αφορά τώρα την προστασία των δεδομένων και τον επόπτη ε, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αυτά θα πρέπει να τα επανεξετάσουμε πριν ψηφίσουμε στην Επιτροπή, γιατί και αυτά είναι σημείο κλειδί. Πριν ολοκληρώσω, να αναφερθώ και στην αρχή προστασίας δεδομένων. Οι αρχές προστασίας δεδομένων είναι κι άλλο επίμαχο θέμα για τους συναδέλφους. Θα πρέπει να με βοηθήσουν και πραγματικά ζητώ τη συνδρομή σας να συντάξουμε ένα κείμενο το οποίο πραγματικά θα είναι χρήσιμο. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο κριτήριο για να καθορίσουμε ποιε είναι οι αρμοδιότητε τη αρχέ και να δούμε αν θα δεχτούμε το μοντέλο του One Stop Shop που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη ενιαία ε, θηρίδας ή αν θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποια άλλη μορφή. Ε, και είναι εύκολο ε, συχνά και συχνά συμβαίνει το Συμβούλιο να έχει διαφορετική θέση από το Κοινοβούλιο, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και λίγο λογικά. Θα πρέπει να μας ενδιαφέρει η συνεκτικότητα και κυρίως ε, σε εμά επαφίεται να δώσουμε μία συγκεκριμένη, σαφή ε, και ε, κοινή πολιτική κατεύθυνση, την οποία θα συμμερίζονται οι περισσότερες πολιτικές ομάδες. Και θα πρέπει να κάνουμε και μία πολιτική επιλογή για τις συμβιβαστικές τροπολογίες που σχετίζονται με τα μέτρα, τις ευθύνες και τις κυρώσεις στην ε, γνωμοδότησή μου είχα επικεντρωθεί αποκλειστικά στη συνάφεια μεταξύ των αποφάσεων των διαφόρων αρχών, αλλά είχα αφήσει στην άκρη το θέμα των κυρώσεων, ε, που θεωρούσα ότι αποτελούν αναστατικό παράδειγμα για τις παραβιάσεις, αλλά οι συνάδελφοι φαίνεται ότι θέλουν να παρέμβουν και στις κυρώσεις και στα ποσοστά ε, τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη. Γι' αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια πρακτική λύση και μια συμβιβαστική λύση. Τώρα για τις πράξεις κατεξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις αυτές τις έχουμε σε όλο τον κανονισμό. Ε, παρακολούθησα τις εργασίες της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και εκεί γίνεται και μια μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να καθαρίσουμε ποιες είναι οι απαραίτητες, να αντικαταστήσουμε ε, τις άχρηστες και να ε, διαγράψουμε αυτές οι οποίες θεωρούμε ότι είναι περιτές. Θα πρέπει λοιπόν και εδώ εμείς να συνεργαστούμε με όλες τις πολιτικές ομάδες προκειμένου να επιτύχουμε το στόχο μας να έχουμε ε, μια εσωτερική αγορά που θα έχει εναρμόνιση και θα προστατεύει τον καταναλωτή. Προκύπτει λοιπόν ε, μια ανάγκη να τηρήσουμε τα όσα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρά το γεγονός ότι ορισμένα πράγματα θα πρέπει να είναι ε, πρωτίστως πολιτικού χαρακτήρα. Υπάρχει λοιπόν μια καλή βάση ε, συνεργασίας αλλά ακόμα δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την πλήρη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γι' αυτό και ακριβώς στις διάφορες επιτροπές προσπαθούμε να καθορίσουμε μια σειρά από συμβιβαστικές προτάσεις και τροποβελτιώσουμε αυτόν τον κανονισμό. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους συναδέλφους για την ε, προθυμία τους να συνεργαστούν και για το γεγονός ότι είναι διατεθειμένοι να συνεισφέρουν στις συμβαστικές προτάσεις, οι οποίες θα είναι ουσιώδεις διότι παρά το γεγονό ότι η δική μα είναι απλώ μια γνωμοδότηση, είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο μα και καθοριστική σημασία ε, και για την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Σα ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σα για σχόλια. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Κόμη. Όλοι συμφωνούμε μαζί σας για τη σημασία του έργου αυτού που θα βοηθήσει την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να προχωρήσει με μια πρακτική και αποτελεσματική πρόταση. Προχωρούμε στους κοιόδης και να σας πω ποιοι είναι και στον κατάλογο των ομιλητών. Uh, Αυτή είναι η ισχυώδης, ε, ο κύριος Κάλλο, ο κύριος Χέντ, και ο κύριος Στάιλος επίσης. Η κυρία Σαλδεμόζε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Κόμη για την πολύ καλή παρουσίαση. Ευχαριστούμε για την πολύ καλή παρουσίαση που δείχνει το ενδιαφέρον για την προστασία των δεδομένων. Δείχνει και τη σημασία της πρότασης αυτής και ότι είναι δύσκολο να εναρμονίσουμε ένα πράγμα όπως η προστασία δεδομένων διαμιάς σε επίπεδο ένωσης. Γιατί, διότι υπάρχουν πολλές μεγάλες πολιτισμικές διαφορές στον τρόπο χειρισμού των δεδομένων και πολλές διαφορετικές παραδόσεις. Είναι πολλές οι τροπολογίες. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται χρόνος για να έχουμε πλήρη εποπτεία πώς θα δώσουμε συνέχεια στο φάκελο αυτό. Και προσβλέπω στην ε, συνάντησή μας με τους Σκιώδης την επόμενη εβδομάδα για να βρούμε κάποιο κοινό έδαφος για να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες. Σήμερα θα μιλήσω λίγο για τις ε, προθέσεις της Ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για την προστασία δεδομένων, τα μέλη της ομάδας μας κατέθεσαν 75 τροπολογίες, όχι τόσες πολλές όσες ε, η συγκήτρια, αλλά η ουσία των προτάσεων μας είναι ότι στηρίζουμε την προσέγγιση της Κομισιόν, θέλουμε ισχυρό κανονισμό που θα υποστηρίζει τους καταναλωτές. Παράλληλα όμως, θέλουμε να υπάρχει περιθώριο ευελιξίας επίσης, όπως ανέφερε άλλωστε και η συγγήτρια. Και πρέπει να προβλέψουμε ευελιξία και στους διάφορους τομείς και στα διάφορα κράτη-μέλη. Ανάλογα είναι κανείς μη κερδοσκοπική οργάνωση, για παράδειγμα, ή κάποια εταιρεία η οποία ε, βγάζει χρήματα από τα δεδομένα των ανθρώπων. Αυτό που θέλουμε στην ομάδα μου είναι, για παράδειγμα, να ενισχυθούν οι προϋποθέσεις της ιδιωτικής σφαίρας ε, έμεσα και διασχεδιασμού. Αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι να επιτρέψουμε στο δημόσιο τομέα να κάνει έρευνα τομεακή και εκεί να χρησιμοποιεί δεδομένα, πάντοτε όμως με βάση την προσέγγιση ότι το δημόσιο, η κοινή γνώμη θα είναι δεδομένη ότι δεν θα γίνεται κατάχρηση των δεδομένων, της χρήσης των δεδομένων. Όταν μιλάμε για μη κυβερδοσκοπικές οργανώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα προσήπουσας χρήσης των δεδομένων. Παράδειγμα, από τη μια πλευρά θα πρέπει να είναι δυνατόν οι εκκλησίες, για παράδειγμα, να κάνουν εράνους για βοήθεια, ανακούφιση κλπ. Αν όμως πει κάποιος ότι εγώ δεν θέλω να με να ε, πλησιάσει άλλη φορά η τάδε οργάνωση γιατί δεν θέλω να κάνω δωρεά, τότε θα πρέπει να είναι βέβαιο ότι οι οργανώσεις θα μπορούν να προστατεύουν το πρόσωπο αυτό για να μην ε, έρθουν σε επαφή άλλη φορά μαζί του. Αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει να μπορούν να αποθηκεύουν τα δεδομένα που λένε ότι δεν πρέπει να, ε, όσο θέλει να ξανάρθουν σε επαφή. Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει μια ευελιξία η οποία θα προστατεύει τους πολίτες και το αντικείμενο των δεδομένων, από την άλλη όμως θα διευκολύνει τις οργανώσεις να χειρίζονται με τον προσήκοντα τρόπο τα δεδομένα. Επίσης είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη μας και τις συλλογικέ συμβάσεις. Ένας εργοδότης θα μπορεί να έχει και τοπικές πολιτικές δεδομένων και δεν ξέρω αν η τωρινή πρόταση το καλύπτει αυτό. Συμφωνούμε με την εισηγήτρια στο θέμα της δημιουργίας προφίλ. Πρέπει να το εξετάσουμε αυτό. Ίσως εκπλήσει, αλλά θέλουμε τους καταναλωτές και ιδιαίτερα τα παιδιά μας να είναι προστατευμένα απέναντι σε αυτό. Όμως ε, υπάρχουν τόσο πολλές τροπολογίες που είναι αδύνατο να τις καλύψουμε τώρα. Πάντως η συνολική μας προσέγγιση είναι ότι θέλουμε ισχυρή οδηγία αλλά και ευέλικτη. Και όλοι όσοι χειρίζονται δεδομένα θα πρέπει να μπορούν να κάνουν ακριβώς αυτό πρέπει να βρούμε και συμβιβαστικές τροπολογίες και περιμένω με ενδιαφέρον τις εργασίες μας τις επόμενες εβδομάδες. Δεν θα είναι εύκολο, το ξέρω, αλλά θα είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ ενδιαφέρον ο φάκελος αυτός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να συγχαρώ Υπάρχουν πολλές τροπολογίες και, και μόλις τελείωσα την εργασία με το φόρουμ του ε, Έρασμου, όπου έχουμε πάνω από χίλιες τροπολογίες, δηλαδή αυτό δεν εντυπωσιάζομαι με αυτές. Εν πάση περιπτώσει είναι πολλές οι τροπολογίες και σημαίνουν σκληρή δουλειά. Προσβλέπω σε αυτό επειδή είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και όπως και οι περισσότεροι από εμά, υπάρχουν πολλές ομάδες ενδιαφερόμενες, πολλές επιχειρήσεις που έχουν πραγματικό συμφέρον και ενδιαφέρον για αυτό το θέμα και χρειάζεται να γίνει σκληρή δουλειά για να βρεθεί σωστή ισορροπία. Και αυτό θα ήθελα να σας πω σήμερα. Εξ ονόματο τη ομάδα ALDE προσπαθώ να βρω ισορροπία μεταξύ των ετοιμάτων των καταναλωτών και των χρηστών αφενό και αφετέρου τη επιχειρήσει που επιθυμούν να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες που τους παρέχουμε εμπορικά. Νομίζω ότι πρέπει να παρατηρούμε τις επιχειρήσεις να ε, χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες και η πρόταση επιτροπής είναι αρκετά προχωρημένη, είναι ευρύτατη, βλέπει στο μέλλον και νομίζω ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί για να βρεθεί σωστή ισορροπία. Αυτό με απασχολεί κυρίως. Ω εκπρόσωπος της ομάδα Άλντε. Πρέπει να είμαστε σωστοί και δίκαιοι όταν μιλάμε για καταστρατήγηση κανόνων. Εάν ανταποκριθεί σε όλες τις προϋποθέσεις μια επιχείρηση, νομίζω ότι δεν μπορούμε να... Είναι ένα πρόβλημα να υπάρχουν μεγάλα πρόστιμα. Γι' αυτό και εκεί πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Υπάρχουν πολλοί τομεί τους οποίου μπορώ να αναφέρω, αλλά επιφυλάσσομαι ε, αναμένοντας την ένταξη των διαπραγματεύσεων, διότι από ό,τι έχω καταλάβει έχουμε προχωρήσει πολύ περισσότερο, περισσότερο από τι άλλε επιτροπέ. Και αυτό οφείλεται ε, στην εισηγήτρια. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίω, όταν ε, συζητήσουμε ευρύτερα το θέμα θα επιστρέψουμε στι λεπτομέρειες. Όπως σας είπα όμως, οι Άλντε πιστεύει ότι πρέπει να βρεθεί ισορροπία ανάμεσα ε, στους καταναλωτές, στους χρήστες του ίντερνετ και τι επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι όπως είπαν όλοι, αυτό το θέμα είναι μεγάλο περίπλοκο. Αλλά έτσι είναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εκεί η εντύπωσή μου είναι ότι βασικά όλοι θέλουμε το ίδιο πράγμα, δηλαδή κάτι το οποίο θα προστατεύει τους πολίτες, αλλά και που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λειτουργούν στην Ευρώπη. Συνεπώς, δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων εδώ, αν θέλετε, ή ιδεολογικών συμφερόντων, μάλλον να βρούμε τον τρόπο για να λειτουργήσει στην πράξη. Νομίζω ότι η συγκεκριά έκανε πολύ καλή δουλειά, εν πωλής, Ας δούμε μερικά θέματα. Πρώτα απ' όλα, ε, η συγγήτρια προσπαθεί να απαλλαγεί από θέματα, να ξεκαθαρίσει δηλαδή τα πράγματα. Υπάρχουν ε, πολλές ε, πράξεις οι οποίες όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει εμείς να αφήσουμε τις ευθύνες μας Εάν τα πράγματα είναι περίπλοκα, θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Δεν θα τα υποβάλουμε έτσι κυρίω τη πράξη κατεξουδότηση στην Επιτροπή. Τώρα, όσον αφορά τι διάφορε τροπολογίε, έχω την εντύπωση ότι έχουμε ένα κοινό προβληματισμό, ότι δηλαδή μπορεί να συγκρουστούμε την ελευθερία της έκφρασης ή με τέτοια θέματα. Η συγγήτρια προτείνει να περιλάβουμε την διατύπωση που έχει στην οδηγία του 95. Όχι το δικαίωμα να λησμονηθεί. εάν πρέπει ε, να υπάρχει αυτό σε σχέση με το δικαίωμα της διαγραφής. Ε, πώς θα δημοσιοποιηθούν τα δεδομένα. Νομίζω είναι παράλογο να ζητήσουμε σε κάπου να διαγράψει όλα τα δεδομένα. Καταρχήν είναι αδύνατο, αλλά και δεν είναι και λογικό. Σε πολλές τροπολογίες το, το θέμα αναφέρεται στα ανώνυμα και σε μη ανώνυμα, επώνυμα δεδομένα. Νομίζω ότι πρέπει να παροτρύνουμε, να δώσουμε κίνητρα σε επιχειρήσεις να αναφέρουν ανώνυμα δεδομένα όταν δεν χρειάζεται να κατονομάσουν από πού προέρχονται τα δεδομένα. Αυτό πρέπει να το δούμε προσεκτικά, προσπαθώντας τα κριτήρια αυτά να γίνουν πιο χαλαρά, στο μέτρο του δυνατού βεβαίως, ώστε να δοθεί αυτό το κίνητο στις επιχειρήσεις. Κατόπιν ε, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων. Εδώ δύο θέματα με απασχολούν. Πρώτα απ' όλα δεν θέλουμε να υπάρχουν υπερβολικοί κανονισμοί. Με κάθε κλικ που κάνει κανεί ε, στον υπολογιστή ε, βρίσκει ένα εικονίδιο και λέει το δέχεστε δεν το δέχεστε. Πρέπει να είμαστε πρακτικοί. Για παράδειγμα, αν θέλω να ε, ζητήσω από το τηλέφωνο τα εστιατόρια, είναι σαφές ότι αν πω το nearby, κοντά τι είναι, μπορεί να μην καταλάβει το τηλέφωνο τι σημαίνει το nearby. Γι' αυτό κάθε φορά όταν ε, χρησιμοποιεί τον υπολογιστή μας ζητούν αν συμφωνούμε ή όχι να κάνουμε κλικ σε ένα εικονίδιο. Αλλά πρέπει να προσέχουμε να μην έχουμε ε, ένα κανονισμό που να επιτρέπει στην επιχείρηση να κάνει οτιδήποτε θέλει εφόσον έχει ένα εικονίδιο ε, στο κομπιούτερ, στον ιστότοπο. Δηλαδή η συγκατάθεση δεν απαιτείται πάντοτε για αυτή την υπηρεσία. Και ίσως δεν πρέπει να αποτελεί μέρος αυτού, διότι μπορεί να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου οι εταιρείε μπορεί να χρησιμοποιήσουν προσωπικά δεδομένα τα οποία δεν είναι χρήσιμα αλλά ε, δεν έχουν άλλη επιλογή. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Επίσης με απασχολεί το 6.1.F, f ε, νόμιμα συμφέροντα του υπευθύνου για την επεξεργασία των δεδομένων. Ποια είναι τα έννομα συμφέροντα ε, της επιχείρησης. Αυτό μπορεί τα ένα μας σημαίνει της να κερδίσω το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Τώρα, για το δικαίωμα να αποκτήσει κανείς μόνο του τις πληροφορίες, νομίζω ότι καλό είναι να συγχωνεύσουμε τους δύο κανονισμούς, διότι υπάρχει το δικαίωμα να αποκτήσει κανείς μόνο του πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου να υπάρχουν σε μια ευανάγνωστη μορφή, αυτό είναι λογικό. Αλλά η τροπολογία που κ. Μακλόκιν ε, πρότεινε για το άρθρο 12.2 είναι λογική. Πληροφορίες πιστώσεων. Δηλαδή, αν μπορεί να αποκτήσει κανείς αυτές τις πληροφορίες, που μπορεί κανείς να τις διαβάσει, θα μπορούσε όμως να δημιουργήσει ατασταλίες και απάτες. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις όπου τα ευαίσθητα δεδομένα δεν θα πρέπει να εμφανίζονται σε μία αναγνώσιμη μορφή από τον καθένα. Αλλά και την αιτιολογική σκέψη 55 και την δικαιολόγηση που δίνει η συγγήτρια αναφέρει ότι αν μπορώ να βγάλω το ιστορικό από μέσα και να το στείλω αλλού. Οι μεγάλες υπηρεσίες δεν πρέπει να διατηρούν τους πελάτες ε, καθαρίζοντας υπηρεσίες, αλλά παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες. Και τέλος το profiling. Από τη μία πλευρά, η κατάρτιση του προφίλ. Μπορεί να κάνουν οτιδήποτε για να μου στείλουν ε, διαφημίσεις. Πολύ καλά, αν επιτύχουν εντάξει, αν δεν επιτύχουν δεν πειράζει. Αλλά από την άλλη πλευρά, Εάν η κατάρτιση προφίλ μπορεί να οδηγήσει σε διάκριση εναντίον κάποιου λόγω της, ε, των σεξουαλικών του προτιμήσεων ή της φιλής του κτλ. Ε, δεν θα πρέπει να το δεχτούμε. Πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός των περιπτώσεων. Όπως είπα όμως, βασικά τα ίδια πράγματα επιζητούμε. Και γι' αυτό προσβλέπω στην συνάντηση των σκιωδών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ένα-δυο σύντομες παρατηρήσεις και θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι σύντομος. Είμαι λοιπόν συνσκιώδης ε, συντάκτης με τον κύριο Μπίλεν λοιπόν. Είναι πολύ σημαντική αυτή η γνωμοδότηση και χαίρομαι που προσπαθούμε να κινηθούμε αυτή τη στιγμή διότι ο, ο κόσμος προσπαθεί να βρει κατευθύνσεις από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών γίνονται πολλά πράγματα, αλλά εμείς έχουμε πολύ καλό ιστορικό, διότι πάντα ε, καταλήγουμε σε ρεαλιστική νομοθεσία. Και πρέπει να σας πω ότι διαδραματίσαμε πολύ σημαντικό ρόλο ε, με την Επιτροπή ε, Πολιτικών Ελευθεριών για την οδηγία η οποία για πρώτη φορά ε, περιλάμβανε ε, στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την κοινοποίηση χρήση δεδομένων. Και αυτό το έχουμε ξεχάσει και ε, με εκπλήσει το γεγονό ότι οι τρέχουσε προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπής δεν αντανακλούν την νομοθεσία που πέρασε η Επιτροπή μα. Όσον αφορά τώρα τις ε, κατεξουσιοδότησης πράξεις που συζητήσαμε και στο παρελθόν και είπε και ο κύριος Έγκστρομ προηγουμένως, θα ήθελα να υπενθυμίσω στην Επιτροπή ότι η αρχική πρόταση που λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οδηγία περιέλαμβανε ε, και μία κατεξουσιοδότηση ευθύνη για όλα όσα αφορούν την πρώτερη κοινοποίηση δεδομένων. Επομένως, εμείς από την Επιτροπή μας είπαμε ότι ήταν απαράδεκτα αυτά και αυτές είναι πολύ σημαντικέ πολιτικές αποφάσεις για τους καταναλωτές και ουσιαστικά εμείς σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων γίνεται η κοινοποίηση της προστασία των δεδομένων. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι διατάξεις και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι εμείς έχουμε ήδη συμφωνήσει για πράγματα προστασίας των δεδομένων και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και προτείνουμε κατά την άποψή μας ε, τροπολογίες που μας ε, κρατούν πιο στενά συνδεδομένους με την αρχική ρεαλιστική προσέγγιση που είχαμε εμείς για την προστασία δεδομένων και όχι αυτά τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι όλοι επιθυμούν μια οδηγία η οποία θα είναι σαφής και ε, νομικά ε, ακριβής και έτσι θα είναι αποτελεσματική. Πρέπει να είναι απλή και σαφής για αυτούς οι οποίοι θα εφαρμόζουν την οδηγία, που ουσιαστικά είναι αυτοί που χρησιμοποιούν για εμπορικούς λόγους δεδομένα, αλλά όπως επίσης είπε ε, και κάποια συνάδελφος, και χρήστες του δημοσίου τομέα, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικά και κάποιες από τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον τρόπο με τον οποίο είναι διατυπωμένες δεν είναι αρκετά σαφείς και δεν επικεντρώνονται στα κρίσιμα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε. Χρειαζόμαστε μία πλήρως εναρμονισμένη οδηγία διότι ε, έτσι θα αντιμετωπίσουμε και την παρούσα κατάσταση στην πραγματικότητα. Ε, αρκετές οργανώσεις σε διάφορες χώρες διατηρούν προσωπικά δεδομένα σε ε, Cloud υπολογιστών ή σε βάσεις δεδομένων αλλού και θα πρέπει να υπάρχουν κοινέ διατάξεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι λοιπόν υπέρ της πλήρους εναρμόνισης. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι σαφές ότι αυτό είναι πολύ σημαντική προϋπόθεση για την Επιτροπή μας, γιατί νομίζω ότι ένα από τα ε, προβλήματα που αντιμετωπίσαμε είναι ότι ναι μεν κάποια κράτη-μέλη κατανοούν ότι υπάρχει ανάγκη για πλήρη, ε, πλήρως εναρμονισμένη πρόταση, αλλά από την άλλη δεν συμφωνούν με τα όσα θέλει να συμπεριλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι διαφωνούν με την πλήρως εναρμονισμένη πρόταση. Πρέπει λοιπόν κατά κάποιο τρόπο να προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο πιο ισορροπημένοι στο πώς θα προχωρήσουμε. Κάτι επιπλέον, τα συμφέροντα και η προστασία των καταναλωτών. Εμείς είμαστε πολύ ευαίσθητοι εδώ στην Επιτροπή μας για το θέμα αυτό και θα ήθελα να επανέλθω στις σημαντικές διατάξεις που συμφωνήσαμε για τη διαφάνεια για τους καταναλωτές, ε, για την περίπτωση των cookies. Θυμάστε τη συζήτηση κάναμε ε, τότε γι' αυτά και ε, το θέμα είναι τι συνάνεση απαιτείται για να γίνει κάτι τέτοιο και ποια είναι η σχέση μεταξύ του να διαβιβάσουμε ένα μήνυμα διαφάνειας και συνένεσης ε, στους καταναλωτές και με το όσο προσπαθούμε να κάνουμε. Και νομίζω ότι καταλήξαμε σε μια ισορροπία και τώρα εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε πολλές χώρες. Ξέρετε ότι έγινε ολόκληρη συζήτηση για το θέμα αυτό. Αλλά ε, είναι πολύ σημαντική η σχέση που υπάρχει εδώ. Αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι στους καταναλωτές εν γέννη αρέσει να κάνουν συναλλαγές στο διαδίκτυο. Αν δείτε, ε, οι online συναλλαγές είναι οι πιο διαδεδομένες και αυτές οι οποίες αυξάνονται περισσότερο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εύκολο και βολικό να κάνει κάποιος συναλλαγές ε, στο διαδίκτυο και μας ενδιαφέρει όμως να υπάρχει εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη είναι ότι όταν δίνουν τα προσωπικά τους δεδομένα, ε, και ξέρουν ότι ε, όταν κάνουν μια συναλλαγή αναπόφευκτα κάποια από αυτά τα στοιχεία θα περάσουν κάπου. Εάν λοιπόν επιτρέπουν σε κάποιον προμηθευτή να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα, ε, θέλουν να είναι σίγουροι ότι τα χρησιμοποιούν με υπεύθυνο τρόπο και ε, δεν θα χρησιμοποιούνται τα δεδομένα για κάτι το οποίο δεν εγκρίνουν. Και αυτό λοιπόν και για λόγους διαφάνειας είναι πολύ σημαντικό. Και ο όλος στόχος αυτής της πρότασης είναι να είναι σαφές στους χρήστες των δεδομένων τι υποχρεώσεις έχουν και πώς πρέπει να τα χρησιμοποιούν από εκεί και πέρα για λόγους διαφάνειας. Και επομένως, πράγματα όπως η κατάρτιση προφίλ που για κάποιους ανθρώπους ε, είναι τμήμα της διαδικασίας η κατάρτιση προφίλ. Παραδείγματο χάρη, αν αγοράσουμε βιβλία, μας κάνουν προσφορές για βιβλία ε, τα οποία είναι αντίστοιχα με τις ε, αρχικές μας επιλογές. Κάποιους δεν τους ενοχλεί αυτό και δεν έχουν καμία ένσταση από αυτού. Η ανεπιθύμητη χρήση του προφίλ τους όμως και το αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας είναι που μπορεί να ενοχλεί και να πρέπει να εξετάσουμε. Αυτά όλα λοιπόν είναι πολύ σημαντικά. Θα πρέπει να προτείνουμε λοιπόν ε, κάποιες τροπολογίες τις οποίες μπορεί εσείς να θεωρείτε δύσκολες, αλλά νομίζω ότι το θέμα εδώ είναι ότι οι καταναλωτές δεν συνειδητοποιούν την αξία και τη σημασία των δεδομένων που, τους αρέσει, ε, που έχουν. Ορισμένες φορές τους αρέσει να χρησιμοποιούν τα δεδομένα τους ε, για κάτι το οποίο θεωρούν σημαντικό, αλλά αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα αυτά είναι πολύτιμα για αυτόν το, ο τα χρησιμοποιεί. Και ε, θα πρέπει να δούμε λοιπόν και τι αξία ε, προσδίδουν οι καταναλωτές στα δεδομένα. Τμήμα της αξίας είναι ότι λαμβάνουν υπηρεσίες, αυτά σχετίζονται και με τη ε, διαφήμιση και νομίζω ότι οι καταναλωτές το κατανοούν αυτό και δεν είναι και απαραίτητο αντίθετοι σε κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα όμως τα ωφέλη τα οποία αποκομίζουν από τα δεδομένα και το πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους, αυτό είναι σημαντικό. Και κάτι τελευταίο, για να μην το λησμονήσουμε και αυτό, για το δικαίωμα διαγραφής ε, του καταναλωτές. Νομίζω ότι η έννοια του δικαιώματος διαγραφής δεν ορίζεται καλά στη συγκεκριμένη νομοθεσία και νομίζω ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων τους. Αλλά το θέμα είναι ε, μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να φτάσουμε ώστε να μην αναιρέσουμε τα συμφέροντα του καταναλωτή. Και δεν θα πρέπει απαροτήτως να θεωρείτε ότι κάποιος θα ζητά να διαγραφεί το ιστορικό του, διότι μπορεί να ε, βοηθήσει και στην προστασία του καταναλωτή. Παραδείγματος χάρη, έστω ότι εσείς πωλείτε ένα αυτοκίνητο και κάποιος θέλει να το αγοράσει και εσείς θέλετε να έχετε το ιστορικό του χρήστη για να δείτε αν είχε κάποιο πρόβλημα το αυτοκίνητο ή αν θα υπάρξει κάποιο μελλοντικό πρόβλημα. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για ένα σπίτι το οποίο πουλάτε ή για τη χρήση εξοπλισμού. Ε, Όλα αυτά λοιπόν για μένα είναι θέμα ισορροπίας και πάλι. Και επειδή στις περιπτώσεις που οι πληροφορίες αυτές ε, θα είναι διάφανες, θα είναι στο δημόσιο χώρο, το αυτοκίνητο αυτό δεν είναι απλώς ε, ιδιοκτησία σας, ε, το να μπορεί κάποιο λοιπόν να επεξεργαστεί αυτά τα ανώνυμα δεδομένα για να δει τι προβλήματα μπορεί να έχει ένα αυτοκίνητο που τυχόν θα πουλήσετε, είναι ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ ότι αυτά θα πρέπει να τα κάνουμε μαζί και ελπίζω ότι αυτά θα αποτελέσουν και προστιθέμενα αξία για τη συζήτηση. Ο κύριος Σαλβίνη νομίζω είναι ο τελευταίο εκ των σχεδόν εισηγητών και μετά θα ακούσουμε του υπολείπου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Τα περισσότερα τα ακούσαμε, επομένω, δεν θα τα επαναλάβω κι εγώ ε, για λόγους οικονομίας χρόνου Καλή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενδιαφέροντα τα όσα έχει να μας πει η συγγήτρια. Δύο-τρία σημεία τα οποία θα ήθελα να επισημάνω. Εμείς ως ομάδα της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας προτείναμε ελάχιστα γιατί θεωρούμε ότι το σημείο κίνησης είναι καλό ω προ τα μέσα κοινωνική δικτύωση, τα οποία εξακολουθούν να αυξάνονται όλο ένα και περισσότερο, χωρί ε, να ψάχνουμε δαίμονες, αλλά για να αναλάβουν τις ευθύνες τους ε, αυτοί οι διεθνείς φορείς, ε, για να προστατεύσουν στρατηγικές ε, και δεδομένα τα οποία αφορούν πλέον εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την διατήρηση των δεδομένων σε τρίτη χώρα διευκρινίζουμε ποια θα πρέπει να είναι η νομοθεσία που θα πρέπει να εφαρμόζεται για κάποιον χρήστη ο οποίος από το Βέλγιο, την Ιταλία ή από κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιεί αμερικανική ιστοσελίδα ή κινέζικη ιστοσελίδα που διατηρεί τα δεδομένα του, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει μόνο η online χρήση. Ε, υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια πολιτών ή καταναλωτών, παρά το γεγονός ότι δεν μ' αρέσει ο όρος. Ε, σκεφτείτε του ηλικιωμένου που δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο κατά βάση, αλλά του καλεί κάποιο στο τηλέφωνο του στο σπίτι για να αγοράσουν κάτι και υπάρχουν ε, εκατοντάδε εταιρείε που διαθέτουν τα στοιχεία του ε, και χωρίς την έγκρισή του. και επομένω, ναι με να επικεντρωθούμε στο διαδίκτυο, αλλά να σκεφτούμε και αυτού του ανθρώπου που δεν ήρθαν ποτέ σε επαφή με το διαδίκτυο και τον υπολογιστή, αλλά αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Να τονίσουμε λοιπόν ότι ε, υπάρχουν και δικαιώματα για τους καταναλωτές αλλά και δικαιώμα ε, για τις επιχειρήσεις. Επομένως, προσπαθούμε λίγο να καθορίσουμε κάποιες λεπτομέρειες. Επικεντρωθήκαμε σε κάποιες από αυτές, ε, όπως για παράδειγμα στο άρθρο 7 για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη με τη μορφή των δεδομένων και τους κινδύνους που ελοχεύουν. Όπως είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής μας, υπάρχουν πιο ευαίσθητες αγορές από άλλες και πιο ευαίσθητα στοιχεία. Καλή δουλειά εύχομαι στην εισηγήτρια και θα πρέπει ως στόχο να ε, μην δώσουμε την εντύπωση ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερη γραφειοκρατία, θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες ευθύνες. Θεωρούμε ότι λίγα είναι αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε, διότι έχουμε πολύ καλό σημείο κίνησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουμε όλε τι συνεισφορέ από τα μέλη. Ξεκινάμε με την κυρία Δασβενή. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω και να χαιρετήσω την παρουσίαση που κάνετε σήμερα και την εξαιρετική γνωμοδότηση δεν έχουμε πολλά να προσθέσουμε, διότι ήταν όλα πολύ κατανοητά. Συμφωνώ και με τα περισσότερα και με του περισσότερου συναδέλφου. Θα ήθελα να προσθέσω τα εξή. Πρώτα απ' όλα, η προστιθέμενη αξία αυτή τη Επιτροπή, όπω υπόθηκε πολύ σωστά, είναι να δημιουργηθεί μια ισορροπία ανάμεσα στη μέγιστη προστασία ε, των καταναλωτών, που είναι το αντικείμενο τη Επιτροπή μα, και τη ενιαία αγορά, σε μια τη στιγμή που παγκόσμια τεχνολογία αναπτύσσεται ταχύτατα και πρέπει να ενισχύσουμε την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας. Συμφωνώ, ακόμα και οι Έλληνες συνάδελφοι είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν μια πραγματιστική, πρακτική προσέγγιση θα ήθελα να μιλήσω για τον κανονισμό και όχι για την οδηγία. Εμείς έχουμε ένα επιπλέον καθήκον να καταστήσουμε τον κανονισμό εφαρμόσιμο αμέσω στον πραγματικό κόσμο, δηλαδή στους καταναλωτές οι οποίοι ε, είναι άτομα ανεξάρτητα, αυτόνομα, με ελεύθερε επιλογές. Και βεβαίω είναι αφιλοκερδής ε, οργάνωση του δημόσιου τομέα που θα πρέπει να σέβεται στους καταναλωτέ. Εδώ ε, ε, ε, στον αγαπητό φίλο Μούσα, θα ήθελα να πω ότι ελπίζω να συμφωνούμε ότι η πλήρη εναρμόνιση είναι ακριβώ ο δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Και το, η πρόκληση του κατακαιρματισμού, όπω λέει ο Μάξιμο, διότι η διάκριση που κάνετε ανάμεσα ε, στην προστασία δεδομένων για τι επιχειρήσει και τι αφιλοκαιρετικέ οργανώσει δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο ε, τα κράτη-μέλη, τους καταναλωτές, ε, τους κατά εκατομμύρια, τα 500 εκατομμύρια καταναλωτών ε, στις χώρες μας. Νομίζω ότι όταν μιλάμε για ευελιξία είμαστε σαφείς. Ευελιξία για μένα δεν είναι οι εθνικές εξαιρέσεις, διότι διαφορετικά υπονομεύουμε το αντικείμενο του έργου μας χρειαζόμαστε απλότητα, σαφήνεια, νομική ασφάλεια. Όπως έλεγε ο Μάρκο, επίσης πρέπει όλοι οι ορισμοί να γίνουν πιο σαφείς. Τι σημαίνει κατάρτιση προφίλ, τι σημαίνει ε, το αντικείμενο, τι είναι, ε, τι είναι το δικαίωμα της συνένεσης, το δικαίωμα να λησμονηθεί κτλ. Ε, πρέπει να πω ότι πρέπει να κατασύσουμε όλα αυτά σαφέστατα. Γι' αυτό η Επιτροπή πρέπει να φροντίσει ότι όλα να είναι ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα. Γι' αυτό ε, υποστηρίζω την τροπολογία 90 και για να είμαι συγκεκριμένη και σαφής, τα δικαιώματα των παιδιών με απασχολούν ιδιαίτερως. Έχετε δίκιο ότι δεν αφορά μόνο το ψηφιακό κόσμο ε, αυτός ο κανονισμός, αλλά τα παιδιά μας απασχολούν κυρίως στον ε, ηλεκτρονικό ψηφιακό κόσμο και κατέθεσα μια τροπολογία για το δικαίωμα της συνένεσης, της συγκατάθεσης. Νομίζω ότι πρέπει να διατηρήσουμε τον ορισμό του ΟΗΕ για το τι είναι παιδί. Δηλαδή κάτω των 18 ετών, διότι αν αλλάξουμε τον ορισμό του ΟΗΕ, τότε θα υπάρχει, θα δημιουργήσουμε σύγχυση. Όπω σε όλο το έργο που έχουμε κάνει στο Κοινοβούλιο, χρησιμοποιούμε αυτόν τον ορισμό του ΟΗΕ. Για να μην υπάρχει σύγχυση. Το άλλο είναι ότι μέχρι την ηλικία των 13 χρειάζεται η συγκατάθεση των γονέων. Μετά από τα 13, από τα 13 στα 18, Μπορείτε να κάνετε μια διαφοροποίηση μεταξύ ε, των παιδιών και των εμφύβων, αλλά το δικαίωμα της συνένεσης, το δικαίωμα του να λησμονηθεί είναι πολύ σημαντικό και για τους εφήβους. Από τα 14 στο 18 οι έφηβοι δεν θα έχουν καμία προστασία. Ελπίζω να συμφωνήσετε, να με υποστηρίξετε στην τροπολογία μου. Επίσης, ε, η τροπολογία μου 220, 299 που έχει σχέση με την κατάρτιση του προφίλ δηλαδή να υπάρχει μία γλώσσα φιλική προς το παιδί. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό και χαίρομαι που και ο Κρίστιαν το είπε. Δηλαδή, να μην χρειάζονται πολλά χαρτιά να συμπληρώνει κανεί άλλα για τα παιδιά, να αισθανθούν ότι δεν τους κοροϊδεύει κανείς, ότι δεν τους εξαπατά κανείς όταν ζητούμε τη συγκατάθεσή τους. Και πρέπει με τον επιχειρησιακό κόσμο να έχουμε διάλογο για να βρούμε την καλύτερη λύση για τα παιδιά, να υπάρχει το δικαίωμα της συγκατάθεσης του παιδιού. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Κυρία Γκάλο, κυρία κυρία Στάιλερ. Ε, ο κύριος Λόκγκαρντ ήθελε να επανέλθει, η κυρία Σάλντε Μόζερ επίσης. Έχουμε χρόνο για ένα γρήγορο γύρο απαντήσεων και η συγγήτρια θα μιλήσει αργότερα. Πρέπει να αφήσουμε χρόνο και για την Κομισιόν. Και θα τελειώσουμε στην ώρα μας ε, για το διάλειμμα. η συντάκτρια της γνωμοδότησης για την νομική επιτροπή. Για να δούμε αν ε, θα είναι παρόμοια η γραμμή πλεύσης της όπως και εδώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Παρεμβαίνω εδώ πράγματι όχι μόνο ως ε, ε, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής σας, αλλά ως εισηγήτρια της Νομικής Επιτροπής και για τις πληροφορίες που θα σας δώσω πρέπει να γνωρίζετε ότι η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών εκπνέει λίγη σήμερα για την ε, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Μία δεύτερη πληροφορία την οποία θα ήθελα να σας δώσω, προτού εξετάσω εντάχει τα αμφιλεγόμενα σημεία αυτού του κειμένου, ότι στα πλαίσια του φόρουμ, το οποίο ψυχώνω εγώ, αλλά υπό την προσωπική μου ιδιότητα, έστειλα μια πρόσκληση στην κυρία Ρέντινγκ, η οποία την δέχθηκε και συνεπώς θα έλθει να συζητήσει με τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους στις 4 Δεκεμβρίου, 12.30 την Τρίτη. Δεν ξέρω ποια αίθουσα θα είναι, αλλά θα τη βρείτε. Θα βρείτε τις πληροφορίες αυτές. Έρχομαι τώρα και θα είμαι σύντομη επειδή πρέπει να το συζητήσω με ταχύτητα, δεν μπορώ να αναπτύξω όλα τα θέματα, ε, δεν θα είμαι εξαντλητική, αλλά θα επανέλθω σε ορισμένα θέματα που αναφέρθηκαν εδώ. Πρώτα απ' όλα, όπως είπε η συγγήτρια και την ευχαριστώ πολύ, θεωρώ ότι όλα ξεκινάνε από τους ορισμούς και συνεπώς θα πρέπει να διευκρινίσουμε ποια είναι τα ανώνυμα δεδομένα και τα δεδομένα με ψευδόνυμο. Δεύτερη παρατήρηση. Πιστεύω ότι πρέπει οπωσδήποτε να διατηρήσουμε ε, την ρητή συγκατάθεση ως βάση της συνθήκης. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα, ουσιαστικό θέμα. Τρίτη παρατήρηση, ένα σημείο από το οποίο επιμένω και εδώ συμφωνώ με τη συνάδελφα Κορατζά για τα παιδιά. Πιστεύω ότι πρέπει να ξαναδούμε την εξαίρεση από τον κανονισμό που περιέχεται στο άρθρο 2 και που αναφέρει ένα φυσικό πρόσωπο με φιλοκερδή σκοπό στα πλαίσια των προσωπικών δραστηριοτήτων του. Αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά και αυτό υπόθηκε ότι με τα κοινωνικά δίκτυα υπό την προσωπική ιδιότητα μπορεί κανείς να αγγίξει ένα περιόριστο ρυθμό ατόμων και είναι ουσιαστικό να ξαναδούμε αυτή την εξαίρεση επειδή για την προστασία των παιδιών ε, είναι πολύ σημαντική όσον αφορά τα κοινωνικά δίκτυα. Τώρα, για ε, το δικαίωμα στην ψηφιακή λύθη, ε, ως νομική ίσως είμαι πιο αυστηρή, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις υποχρεώσεις του υπευθύνου της επεξεργασίας των δεδομένων να ενημερώσει το ενδιαφέρον άτομο τη στιγμή που ζητάει να διαγραφεί, ε, να διαγραφούν τα στοιχεία. Ε, δεν μπορώ τώρα να επισέλθω στις λεπτομέρειες όλων αυτών των θεμάτων. Αναφέρομαι τώρα στο άρθρο 18 και το δικαίωμα par euh, le rapporteur euh, που και Πιστεύω ότι πρέπει να διαγραφεί αυτό το δικαίωμα μεταφοράς, γιατί επειδή υπάρχει ήδη το άρθρο 15 που επιτρέπει την πρόσβαση και μάλιστα μία πρόσβαση που οδηγεί σε ανακοίνωση. Ε, το άρθρο 18 λοιπόν αν αναφέρεται σε αντίγραφο. Θα ήθελα εγώ να μου πείτε ποια είναι η διαφορά μεταξύ αντιγράφου και ανακοίνωσης ε, ή κοινοποίηση. Νομίζω ότι αυτό απλώς δημιουργεί σύγχυση και αυτό, αυτό το δικαίωμα μεταφοράς θα δημιουργήσει περισσότερες νομικές ασάφειες από ότι διευκρινήσεις. Πάλι εντάχει έρχομαι τώρα σε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο να λυθεί στα πλαίσια του κειμένου, οι σχέσεις μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασία και των υπεργολάβων του, ας πούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ περίπλοκο, επειδή μπορεί να υπάρχουν απεριόριστη υπεργολάβη, χωρίς να το γνωρίζουμε. Γι' αυτό το λόγο προσανατολίστηκα προς μία αρχή γενικής ευθύνης, υπευθυνότητας δηλαδή, του υπευθύνου της επεξεργασίας των δεδομένων, δηλαδή ο πολίτης απευθύνεται σε εκείνον τον οποίο γνωρίζει. Και προβλέπω το εξής, αν αυτό το άτομο δεν είναι το υπεύθυνο της ε, παράβασης, τότε εκείνος θα στραφεί κατά του άλλου επαγγελματία, ο οποίος θα είναι ο υπεύθυνο, αλλά δεν θα πρέπει ο πολίτης να αναζητήσει τον υπεύθυνο για την καταστρατήγηση. Δηλαδή, ε, στο γαλλικό δίκαιο τουλάχιστον, αυτή είναι μια αρχή που υπάρχει και φαντάζομαι και στις άλλες νομοθεσίες υπάρχει αυτή η αρχή. Νομίζω ότι επίσης πρέπει να διευκρινίσουμε την αρχή της προστασίας των δεδομένων by default. Αυτό είναι το άρθρο 23 παράγραφος 2 που επίσης έχει, κάνει να χυθεί πολύ μελάνη Έρχομαι στο άρθρο 31, δηλαδή η κοινοποίηση ε, στις αρχές ε, που κάνουν τον έλεγχο, πάλι για να μην επιβάλλουμε επιπλέον και δυσανάλογες υποχρεώσεις επιχειρήσεις. Αυτή η κοινοποίηση θα πρέπει να γίνεται, πιστεύω, μόνον σε περίπτωση καταστρατήσεις παράβασης, η οποία επηρεάζει σημαντικά τα ενδιαφερόμενα άτομα. Και έχω εμφιβολίες σχετικά ε, με την προθεσμία των 24 ωρών, προβλέπετε και νομίζω ότι δεν είμαι η μόνη άλλωστε. Προχωράω γρήγορα πάλι, έρχομαι στο άρθρο 51. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτό το τομέα να υπάρχει ένα συνομιλητής μόνον, αλλά δεν πρέπει οι εθνικές αρχές να γίνουν ταχυδρομικά κουτιά. Γι' αυτό το λόγο ε, ζητώ συνεργασία μεταξύ των ε, αρχών ελέγχου. Επίσης είμαι υπέρ τη ανεξαρτησία τους, κυρίως ε, στην εκτίμηση των διοικητικών κυρώσεων που θα επιβληθούν και α ε, καθοριστούν ορισμένα επίπεδα, όρια και όπω πολλοί συνάδελφοι, τελειώνω, τελειώνω πρόεδρε, όπω πολλοί συνάδελφοι θεωρώ ότι υπάρχουν υπερβολικά πολλές πράξεις ε, κατεξουσιοδότηση και θα μπορούσαμε να τις περιορίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όπως είπαν και άλλοι, ο στόχος του νέου κανονισμού είναι η επαρκής προστασία των καταναλωτών. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι επιφυλακτική σε σχέση με, την καταρχήν, ε, με τον καταρχήν αποκλεισμό, την εξαίρεση των ε, μικρών επιχειρήσεων από τον κανονισμό, γιατί έτσι υποβαθμίζεται η ποιότητα της προστασίας. Γιατί πόσες επιχειρήσεις ενδεχομένως θα κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας. Δηλαδή αυτοί που έχουν κάτω από 250 εργαζομένους μπορεί να θίγονται εδώ, ενώ πρέπει να συμμετέχουν και να συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις. Συνολική προστασία πρέπει να παρέχεται. Χρειάζεται σαφής προστασία, πληροφόρηση στους καταναλωτές που πρέπει να ξέρουν τι πληροφορίες λέγονται τι χρησιμοποιούνται. Και οι επιχειρήσεις έχουν την ευθύνη να είναι όσο γίνεται πιο ασφαλές το σύστημα για να ε, ε, διαφυλάσσεται η ανωνυμία και να ξέρουν οι καταναλωτές ότι είναι προστατευμένα τα δεδομένα τους και θα πρέπει να συλλέγονται και να, διαδίδο, μετα, να διαβιβάζονται όσο γίνεται λιγότερα δεδομένα. Σε ό,τι αφορά τη συλλογή των δεδομένων και το σύστημα, αυτό είναι περίπλοκο και χρήζει περαιτέρω συζητήσεων. Πολύ σημαντικό είναι, όπως ανέφεραν και άλλοι ομιλητές, ε, πολύ σημαντικό είναι το θέμα των παιδιών και των ανηλίκων εδώ πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί και να ισχύουν ιδιαίτεροι κανόνες. Δεν πρέπει δηλαδή να παρεκκλίνουμε εδώ από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Εγώ υποστηρίζω την τροπολογία για την προστασία των δεδομένων σε αντίθεση με άλλα ένομα ε, κοινωνικά συμφέροντα ε, έναντι άλλων συμφερόντων και το άρθρο 6 που ρυθμίζει την διαχείριση των δεδομένων. Δεν είναι δυνατόν ε, τρίτη να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά. Για κανένα λόγο. Επίσης η ε, καταχωρισμένη έρευνα, έρευνα για τον καρκίνο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ή η ενότητα των συλλογικών συμβάσεων είναι σχετικά παραδείγματα. Τώρα για, την, για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις δεν έχω καταθέσει τροπολογίες, αλλά είμαι επιφυλακτική σε σχέση με το να συμπεριληφθούν στην ε, ε, οδηγία θα πρέπει να διευκρινιστεί περισσότερο το θέμα των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να ε, παγρυπνούμε ούτω ώστε να μην ξεπεραστεί κάποιο ελάχιστο πρότυπο. Ε, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα που δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Στάνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια και του σκιώδης. Δεν ξέρω, θα γίνει ακρόαση πάνω σε αυτό το θέμα. Υπάρχει τέτοια προοπτική. Καταλαβαίνω τη συνθετότητα και τον εξισορροπητικό μας ρόλο και ότι πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά. Αυτό είναι σημαντικό γιατί τα δεδομένα είναι ένα θέμα το οποίο θα αναβαθμιστεί σε σπουδαιότητα επειδή ε, τώρα έχουμε και λογαριασμό στο Twitter, όπως μας είπατε, είναι ενδιαφέρον όταν μιλάμε για δεδομένα Εγώ πήρα ένα tweet από ένα φίλο σήμερα, στον οποίο προσφέρθηκαν κάποιες ιδέες χριστουγεννιάτικες και αντικείμενα επιχειρηματικά βιβλία, ε, βιβλία, πολιτικές ε, βιογραφίες, ε, ημερολόγια αθλητικά για εκείνον και για, ημερολόγια για ζωάκια, για την γυναίκα, για χειροτεχνίες, βιβλία, μυθιστορήματα. Υπάρχουν 65 retweet εδώ για το σεξισμό και 150 περίπου favorite παρόλο που ε, είναι ένα θέμα γενικευμένο. Ε, αναφέρουν ε, επίσης διάφορα, διάφορες αστείες απαντήσεις που απορρίπτουν την ιδέα των δώρων. όλα αυτά είναι ενδιαφέροντα και στα κοινωνικά μέσα, αλλά είναι και σημαντικό σε σχέση με το τι πληροφορίες υπάρχουν για μας και πώς χρησιμοποιούνται η Amazon πούμε, πρέπει να μάθουν λίγο για το πώς λανσάρει και κάποια προϊόντα και πώς τα βάζει στην αγορά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και ήθελα να τα πω κάποια στιγμή που δεν, επειδή δεν ήμουν το πρωί. Είστε το πρώτο μέλος της Επιτροπής που χρησιμοποιεί τόσο δραστήρια τα Twitter. Ε, κάποιοι δεν ακούσατε την πρωινή μου ε, ανακοίνωση ότι τώρα έχουμε ένα ε, λογαριασμό στο Twitter. Θα το αναφέρω και στο τέλος, γιατί κάπου τα έχω, τα έχω γράψει τα στοιχεία. Ευχαριστώ. Ναι, ξαναγυρίζουμε σε αυτό που είπα, ότι ναι, η Amazon θα πρέπει να, κάνει, ε, να διαθέσει τις πληροφορίες ε, που έχει για το προφίλ λοιπά. Και αν τις θέλετε μπορείτε να τις διαγράψετε εντελώς. Αυτό έχει να κάνει με τον έλεγχο. Τον έλεγχο και τη διαφάνεια. Δύο σκιώδεις ήθελαν να απαντήσουν γρήγορα και νομίζω η Λάρα Κόμη θα με ενδιαφέρον θα τους ακούσει και θα προλάβουμε και με την Κομισιόν να τελειώσουμε στις 12.30. Ο κύριος Λόκεγκαρτ και μετά η κυρία Σαλντεμόζερ. να απαντήσουν σύντομα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, μια σύντομη παρατήρηση σε αυτά που ακούσαμε. Ε, είναι πολύ σημαντικό και πράγματι ισχύει ότι πρέπει να κάνουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη εναρμόνιση εμείς θα είμαστε υπέρ προφανώς. Από την άλλη, όπως είπα, πρέπει να βρούμε ισορροπία και εν προκειμένου νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ ιδιωτικών εταιριών και δημοσίων εταιριών, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, γιατί κάποια κράτη-μέλη έχουν πολύ προχωρημένο δημοσίο τομέα σε ό,τι αφορά την προστασία συλλογής και προστασίας δεδομένων και σίγουρα δεν θέλουμε να σπάσουμε το σύστημα όταν λειτουργεί. Δεν θέλουμε να καταργήσουμε κάτι το οποίο είναι καταξιωμένο. Όταν κάνουμε τις τροποποιήσεις μπορούμε να την κάνουμε τη συζήτηση αυτή, γιατί αυτός είναι ένας ευέλικτος τρόπος για να προχωρήσουμε, χωρίς να καταστρέψουμε δηλαδή την πλήρη ανωνυμοποίηση, γιατί έχετε δίκιο όταν μιλάω σε εταιρείε, είτε είναι δανέζικες ή διεθνείς εταιρείε φαίνεται ότι έχουν τις ίδιες ιδέες σχετικά με το πώς θα προχωρήσουν στο μέλλον και σίγουρα δεν ε, χρειάζονται σε αυτή την περίπτωση εθνικά συστήματα. Σύνθετο το θέμα, αλλά μπορούμε νομίζω να βρούμε μια συμφωνία. Σας ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Σαλντεμόζε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Λόκεγκαρτ με διευκόλυνε, γιατί και εγώ αυτό προσπαθούσα να πω και ίσως δεν τα κατάφερα. Όταν μιλώ για ευελιξία, νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι στο δημόσιο τομέα έχουμε μια διαφορετική κουλτούρα και διαφορετικές παραδόσεις ε, όταν πρόκειται για το χειρισμό δεδομένων των πολιτών. Πρέπει να γίνουν σεβαστά αυτά κατά κάποιο τρόπο. Αλλιώς ε, θα θυμώσουν οι φορολογούμενοι, διότι στη Δανία και τη Σουηδία, για παράδειγμα, θα πρέπει να φτιάξουμε ένα τελώς καινούριο δημόσιο τομέα για να αντιμετωπίζουν τα δεδομένα. Στις επιχειρήσεις, συμφωνώ, πρέπει να ισχύσει η ενιαία αγορά και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, τα προβλήματα των εταιριών, αλλά πάλι με τρόπο που θα διασφαλίζει ότι θα προστατεύονται καλά οι καταναλωτές. Ναι, στη διαφοροποίηση λοιπόν μεταξύ του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Ήταν εξαιρετική η συζήτηση, πολλά ακούσαμε και τώρα η Κομισιόν θα κάνει κάποιες πρώτες παρατηρήσεις. Ξέρω ότι θα συμμετέχετε και στις μελλοντικέ μας ε, συναντήσεις. Η κυρία Μπολοντζέ θα μας πει κάποια προκαταρκτικά και μετά θα δώσω το λόγο στην κυρία Κόμη για να κλείσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να αντιδράσω. Πρώτα απ' όλα από πλευρά της Επιτροπής ε, βλέπουμε τη γρήγορη εργασία, το έργο που έχει επιτελεστεί την ταχύτητα με την οποία λειτουργήσατε και χαιρετίζουμε όλα αυτά τα γεγονότα. Θα ήθελα να κάνω τις εξής παρατηρήσεις στο παρόν στάδιο, λέγοντας ότι στα διάφορα σημεία τα οποία από την αντικείμενο των τροπολογιών υπάρχουν ορισμένα θέματα ουσιαστικά που αφορούν τη λογική της οικοδόμησης και αρχιτεκτονικής που προτείνεται από την Επιτροπή. Το επίπεδο προστασίας του κανονισμού είναι κανονισμός και το τονίζω, θα πρέπει να σέβεται τη λογική του επίπεδου προστασία που περιέχεται στη σημερινή οδηγία, είτε προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, είτε τη ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων. Ένα βασικό στόχο ήταν να ενισχυθούν αυτέ οι δύο διαστάσει. Από τη μία πλευρά η ενίσχυση των δικαιωμάτων και αφετέρου η διασφάλιση τη καλύτερη λειτουργία στα πλαίσια τη εσωτερική αγορά. Ε, Επίση, προσθέτω ότι ένα νομικό πλαίσιο σαφέ ένα νομικό πλαίσιο εναρμονισμένο, το οποίο θα παρέχει ενισχυμένα δικαιώματα, είναι ένας φορέας ανάπτυξης, ένα στοιχείο εμπιστοσύνη σημαντικό για την καινοτομία και ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Θα ήθελα να επανέλθω σε ορισμένα συγκεκριμένα σημεία ως προς ε, το διοικητικό βάρος. Η πρόταση επιτροπή και σαν αντικείμενο να μειωθεί αυτό το βάρος, το διοικητικό βάρος και γι' αυτό αλλάξαμε όλα αυτά τα συστήματα ε, δύσκολης κοινοποίησης με πιο ευέλικτα συστήματα προσαρμοσμένα στην σημερινή τεχνολογία. Από πλευράς Επιτροπής όμως είμαστε έτοιμοι ε, να βρούμε πώς θα μειώσουμε το διοικητικό άχθο εφόσον βεβαίω η προστασία ε, των δικαιωμάτων των ατόμων δεν πρόκειται ε, να θυγεί. Γι' αυτό θα θέλαμε να συνεργαστούμε. Αναφορικά τώρα με τα σχέδια τροπολογιών που αφορούν βασικές έννοιες. Από πλευράς Επιτροπής πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό πράγματι, υπόθηκε από πολλούς, να έχουμε ένα σαφές νομικό πλαίσιο και είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με τους νομοθέτες για να έχουμε ένα σαφές νομικό πλαίσιο, το οποίο να είναι και εφαρμόσιμο. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια, ε, ένας ευρύς ορισμός της έννοιας των προσωπικών δεδομένων που θα διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων, αλλά επίσης και ε, τις διάφορες υποχρεώσεις που έχουν σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων. Σε αυτά τα πλαίσια η πρόταση της Επιτροπής έχει ένα άρθρο, το άρθρο 10, το οποίο προβλέπει τη διασφάλιση ότι παρά την ευρύτητα των ορισμών δεν θα οδηγούν ε, σε υπερβολικό βάρος στην υλοποίηση των ε, διατάξεων. Τώρα, ω προ τον ορισμό των ανωνύμων δεδομένων και δεδομένων με ψευδόνυμα, αυτά οι έννοιε είναι ενδιαφέρουσε και είμαστε στη διάθεσή σα να τα επεξεργαστούμε στα πλαίσια που ανέφερα, δηλαδή μια προστασία ευρεία και γνωρίζοντα ότι εξ ορισμού τα ανώνυμα δεδομένα δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο ε, προστασίας και δεν καλύπτονται από την πρόταση κανονισμού. Ως προς τις διάφορες τροπολογίες που αφορούν ε, την εδαφική δικαιοδοσία, αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή να έχουμε ένα ουσιαστικό κριτήριο, ένα ε, κριτήριο σαφές και κατόπιν να εξασφαλίσουμε ότι διάφοροι οικονομικοί φορείς ε, να λειτουργούν ίσης όρης. Δηλαδή, φορείς που βρίσκονται εκτός της επικράτησης Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά που έχουν ε, βλέψει στην ευρωπαϊκή αγορά, να μην αντιμετωπίζονται με διαφορετικούς κανόνες όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων. Ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό και που πηγάζει από διάφορε τροπολογίε είναι ότι πιστεύουμε ότι πρέπει στα πλαίσια του κανονισμού να φροντίσουμε να ε, διατηρήσουμε τον ουδέτερο τεχνολογικό χαρακτήρα. Όλα λοιπόν θα πρέπει να ε, έχουν υπόψη, θα, υπάρχουν μελλοντικέ τεχνολογικές εξελίξεις, λαμβάνοντας υπόψη τι θα σημεί σε πέντε χρόνια. Και βεβαίω σήμερα ε, δεν, ε, δεν μπορούσαμε να είχαμε προβλέψει ποια θα ήταν η σημερινή τεχνολογική πρόοδο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στη μελλοντική τεχνολογική πρόοδο. Ένα άλλο που υπόθηκε συχνά είναι το θέμα τη συγκατάθεση. Η συνένεση. Η πρότασή μα ήταν να υπάρχει μία συνένεση, μία συγκατάθεση, καλή όμω συγκατάθεση. Γι' αυτό το λόγο προτάθηκαν πολλά για να ενισχυθεί η ποιότητα τη συγκατάθεση. Βεβαίω όμω συμφωνούμε ότι δεν είναι αναγκαίο να περιορίσουμε, ε, να περιορίσουμε την, δυνατότητα να λειτουργήσει η κοινωνία της πληροφορικής και δεν θέλουμε συνέχεια να κάνουμε κλικ σε τετραγωνίδια και να περιορίζουμε την ε, δυνατότητα αλληλεπίδρασης η συγκατάθεση του ατόμου δεν είναι το μόνο, ο μόνος νομιμότητας. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες νομιμότητας που επιτρέπουν επεξεργασία δεδομένων. Η σύμβαση, η συμβατική σχέση είναι ένας παράγον και ένας άλλος παράγοντας που είναι η ισορροπία των συμφερόντων. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ότι η ελευθερία ε, του επιχειρήν είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο, αλλά το, τα συμφέροντα των ατόμων ή μάλλον ο τρόπο με τον οποίο ε, τα συμφέροντα γίνονται σεβαστά στα πλαίσια τη ελευθερία επιχειρήν μια επιχείρηση η οποία αναπτύσσει τι δραστηριότητέ τη, τα διάφορα στοιχεία πρέπει να επιτρέπουν να υπάρχει ισορροπία και σεβασμό ε, του ατόμου. Συνεπώ, η συγκατάθεση είναι ένα θετικό στοιχείο, αλλά δεν είναι η μόνη δυνατότητα επεξεργασία δεδομένων. Όσον αφορά το θέμα τη ε, κύριας έδρας εγκατάστασης πρέπει να διασφαλίσουμε την ε, νομική ασφάλεια σε αυτά τα πλαίσια και την ενιαία θηρίδα. Επίσης, να υπάρχει μια αρμόδια αρχή με σαφή κριτήρια. Είμαστε διατεθειμένοι να συνδράμουμε για τη διευκρίνηση αυτής της έννοιας, αλλά για την ενιαία θηρίδα ε, πρέπει να έχουμε γνώμονα την απλούστευση και αυτό το στοιχείο της απλούστευσης πρέπει να παραμείνει στην αρχιτεκτονική μας. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι ο πολίτης βρίσκεται μπροστά σε ε, μια θηρίδα ε, εθνικού επίπεδου. Θα πρέπει να έχει ως ε, συνομιλητή τον καταναλωτή σε εθνικό επίπεδο και γι' αυτό θα πρέπει να έχει πολλά μέσα στη διάθεσή του, μηχανισμούς, διάφορες υποχρεώσει. Πρέπει να διασφαλιστεί ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της διευκόλυνσης ε, των επιχειρήσεων αλλά πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η απλούστευση, να υπάρχει μία ενιαία θηρίδα και δεν πρέπει επιχειρήσει να απευθύνονται σε 27 εθνικού ρυθμιστέ, ρυθμιστικέ αρχέ για να λειτουργήσουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Δεν θα μακρηγορήσω για την, τα παιδιά τώρα και την παρέμβαση που έγινε που έλεγε ότι είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε την προστασία των παιδιών μεταξύ 13 και 18 ετών. Η έφηβη e είναι ένας πληθυσμός που πρέπει να προστατευτεί. Κυρίως όσον αφορά το δικαίωμα της λύθης, η, τα παιδιά μεταξύ 13 και 18 ετών θα πρέπει να απολαμβάνουν προστασίες στα πλαίσια ενός βασικού κανονισμού σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν τα Ηνωμένα μια τελευταία παρατήρηση, για να μην περάσουμε το χρόνο μας, ήταν η διάκριση μεταξύ του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα. Εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω πολλά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα το γεγονό ότι η σημερινή οδηγία δεν προβλέπει διάκριση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου υπάρχουν όλο και περισσότερε εταιρικέ σχέσει μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και είναι σημαντικό ε, και οι δύο τομεί να συνεργάζονται με συνοχή, με βάση τι ίδιε αρχέ, εάν ε, θέλουμε να βρούμε ευελιξία, θα τη βρούμε μέσα στον κανονισμό. Η πρότασή μας περιέχει πολλά στοιχεία που διασφαλίζουν ε, ότι θα ληφθεί υπόψη η πραγματικότητα του δημόσιου τομέα στα κράτη-μέλη και είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με εσά για να ληφθεί υπόψη η πραγματικότητα του δημόσιου τομέα στα κράτη-μέλη. Επιμένω όμω ότι σημαντικό είναι να διατηρηθεί η διάσταση της εσωτερικής αγοράς και να εξασφαλίσουμε ότι όλα λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής αγοράς επειδή η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι ένας παράγων ουσιαστικός. Τελευταία παρατήρηση για, το τομέα, για τους τομείς. Όσον αφορά τις πράξεις κατεξουσιοδότηση, η Επιτροπή προβλέπει αυτές τις πράξεις κατεξουσιοδότηση για να Υπάρχει δυνατότητα να εξελιχθούν σύμφωνα με τις νέες τεχνολογίες, να προσαρμοστούν στην τεχνολογική εξέλιξη και να λαμβάνει υπόψη ο γνώμων της εσωτερικής αγοράς. Βεβαίως, ακούσαμε τις ανησυχίες σας και είμαστε διατεθειμένοι να ξαναδούμε ξεχωριστά αυτές τις πράξεις κατεξοδότηση για να δούμε κατά πόσο είναι απαραίτητες και να συνεργαστούμε με τους συνομοθέτες, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν και άλλα μέσα που δεν παρέχουν ίσως το ίδιο επίπεδο νομικής ασφάλειας, αλλά που επιτρέπουν εξειδίκευση. Υπάρχει αυτό που ονομάζουμε checks and balances, έλεγχη και ισορροπία, να δούμε την ενέργεια μεταξύ των στοιχείων και η Επιτροπή είχε προτείνει να δώσουμε μια μεγάλη ε, θέση στον κώδικα συμπεριφοράς που είναι πυλώνας και να υπάρχει ένας μηχανισμός που θα δίνει νομική ασφάλεια και αφετέρου το board, το συμβούλιο που θα περιλαμβάνει όλες τις αρχές προστασίας δεδομένων να καθοδηγεί σε ορισμένους τομείς. Σταματώ εδώ. Ευχαριστώ πολύ διότι μας καθορίσατε κάποια από τα ζητήματα. Θα συνεργαστούμε φυσικά και στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία. Κύριε Κόμη, έχετε κάποιες ε, τελικές παρατηρήσεις να κάνετε για το χρονοδιάγραμμα, για τις προθεσμίες ή οτιδήποτε άλλο. Λάρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, τηλεγραφικά. Λυπάμαι για την ακρόαση, αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Μάλιστα χρειάστηκε να ζητήσουμε από τις υπηρεσίες να καθυστερήσουν κάποιες ε, ημερομηνίε, γιατί η Επιτροπή ΙΜΚΟ είναι από τι πρώτε που θα ψηφίσει. Θα γίνει μια μικρή ακρόαση, ε, μια μισή ώρα στην Επιτροπή Βιομηχανία και Έρευνα. Αν σα ενδιαφέρει, θα μπορούσατε να πάτε εκεί. Εγώ σημείωσα τις διάφορες παρατηρήσεις. Ε, διαπιστώνω ότι σε γενικές γραμμές υπάρχει μια κοινή κατεύθυνση. Στις τροπολογίες θα δοθούν οι καλύτερες κατευθύνσεις. Όσον αφορά τώρα τις προθεσμίες και τα χρονοδιαγράμματα, Εξέταση των συμβιβαστικών τροπολογιών 17 και 18 Δεκεμβρίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή στις 24 Ιανουαρίου. Επομένως, θα πρέπει να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να πιεστούμε λίγο. Ε, θεωρώ ότι η ομάδα δουλεύει καλά, διότι με αρκετούς από τους κοιόδης εισηγητές έχουμε κάνει τόσες πολλές ε, κοινέ εκθέσεις που πλέον ε, καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον στο φτερό. Ε, είναι εξαιρετικό αυτό το εργαλείο, εξαιρετική μέθοδος εργασίας. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν όλους. Για τους ανηλίκους ε, συμφωνώ απολύτως, έχω την ίδια άποψη και εγώ, θα πρέπει να επαληθεύεται και η ηλικία, διότι αυτά είναι από τα βασικά σημεία. Η διάκριση μεταξύ ανηλίκου ε, που φτάνουμε ορισμένες φορές στα 14 με 16 χρόνια και η διαφορά που υπάρχει στον ορισμό του ανηλίκου στις διάφορες χώρες είναι σημαντικό. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι φτάσαμε στις 12.30 ακριβώς με τα όσα σας είπα. Στην ώρα μου κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Επιβεβαιώνω λοιπόν ψηφοφορία στις 24 Ιανουαρίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Και για να απαντήσω και στο της κυρίας ε, Τάιλερ, όντως ε, Υπάρχει ακρόαση προγραμματισμένη για την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ε, και θα υπάρξει και επιτροπή στην, ε, ε, συγγνώμη, ακρόαση στην Επιτροπή Ήτρε. Ελπίζω να μπορέσουμε λοιπόν να μιλήσουμε εκεί. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε στις 3. Συζήτηση για το πώς έχει κατάσταση η οδηγία για τις, στην οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες και σας ανακοινώνω και πάλι τη διεύθυνσή μας στο Twitter.